Good Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας, λέει ο Πρόεδρος και καλώς ήλθατε. Σας παρακαλώ να βάλετε τις ε, κάρτες ψηφοφορίας στην ε, σχισμή. Αρχίζει η ψηφοφορία. Και την κλείνω αμέσω γιατί ήταν δοκιμαστική. Δεν είσαστε και πολλοί, αλλά λειτουργεί πάντως το σύστημα όπως πρέπει. Ας πάμε στην πρώτη ψηφοφορία. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επισήμανση των ελαστικών. Η είναι ο κύριος Μίχαλ Μπόνι. Συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4. Υπέρ, κατά. Ας, ας επαληθεύσουμε. Πρόκειται για την 4 λοιπόν. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται λοιπόν, όπως βλέπετε, συμβαστική 5 υπέρ, κατά, ας επαληθεύσουμε πάλι. Πέρα της ε, ψηφοφορίας. Απερίφθη αυτή. 5α υπέρ, κατά. Α, ας επαληθεύσουμε. 5α, Πέρας. Απερίφθη. Καλά λοιπόν. Ας προχωρήσουμε. Ε, 11 υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε και πάλι. Εννοείται ηλεκτρονικά. Πέρασε. και αυτή. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Και σας παρακαλώ να σηκώνετε καλά τα χέρια σας, γιατί κάπως δύσκολο αλλιώς να μαντέψω τι ψηφίζετε. 81 λοιπόν. Πέρας. Απερίφθηκε αυτή. 80 υπέρ. Κατά αποχές, επαλήθευση. Τέλος. Απερίφθηκε αυτή. 12 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση και πάλι. 12. Τέλος. Απόρριψη. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Τέλος. Απόρριψη. 84 υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε καλύτερα. 84. Τέλος. Απόρριψη. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Πέρας. Απόρριψη. Συμβιβαστική υπαριθμών 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Συμβαστική 10. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. 101 λέει ο πρόεδρος. 101. Υπέρ, κατά, επαλήθευση. 101. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. 112 υπέρ, Κατά. Ας επαληθεύσουμε. Πέρας. Απερίφθη. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση της συμβαστικής έστω και μου φαίνεται ότι απερίφθη μάλλον, Πέρασε. απερίφθη πράγματι. Είκοσι ένα, είκοσι ένα, υπέρ. Κατά, αποχές, Επαλήθευση. Δεν είναι σαφές. Επαλήθευση λοιπόν. 21. Πέρας. 21 ξαναλέω. Εγκρίνεται. 113 υπέρ. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Αυτή καταπίπτει. 13 λοιπόν, συμβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά. Ξαναλέω 140 και κάνουμε επαλήθευση. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά. Ας επαληθεύσουμε. 29 λοιπόν. Τέλος. Απερίφθη. Ενβι 1 υπέρ. Κατά. Α... καλύτερα. NV1. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά Ας επαληθεύσουμε για να είμαστε σίγουροι. Τριάντα εννέα, ξαναλέω. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. 43. Πέρας. Απεριφθεί. 46, 47, 45 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές. Ας επαληθεύσουμε. 4, 46, 47, 45. Τέλος. Εγκρίνονται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε. Την παριθμόν 50. Τέλος. απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. 51. Πέρας. Απερίφθη. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση και σε αυτήν. Τέλος. Απόρριψη. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία επί του σχεδίου όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονικό τρόπο αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. Και συγχαρητήρια στον κύριο εισηγητή. Τώρα, η επόμενη έκθεση πρόκειται για την πρόταση σύσταση Ευρωπαϊκού Βιομηχανικού Τεχνολογικού λοιπά Ευρωπαϊκού Κέντρου Εκανοτήτων. Τώρα, συμβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε. Εδώ ζητείται ονομαστική ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία από την αρχή, συμβαστική 5. Κλείνει. Απερίφθη. Συμβαστική 6. Ονομαστική ψηφοφορία πάλι προβλέπετε εδώ. Τέλος. Εγκρίνεται αυτή. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 273 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13, συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές. Α, εδώ χρειάζεται επαλήθευση. Τέλος. Εγκρίνεται όπως βλέπετε. Καλά λοιπόν. 15 συμβαστική υπέρ κατά αποχές επαλήθευση, διότι συμβαστική είναι. 15. Ε. Εγκρίνεται λοιπόν, μάλιστα. Θαυμάσιο αποτέλεσμα. Συμβαστική 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Τέλος. Κλείνω την ε, ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 21 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται.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 ο πρόεδρο τα είπε λίγο πολύ γρήγορα. Με συγχωρείτε. 29, 29, ε, σωστά. Υπέρ λοιπόν, κατά απόχέ εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά απόχέ εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ, κατά απόχέ, εγκρίνεται. 1, 1, 5, 115 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ, κατά Ας επαληθεύσουμε. Πέρας. Απερίφθη. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3 της ΙΜΚΟ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική σε. Άρα σε παληθεύσουμε καλύτερα. Συμβαστική σι. Εγκρίνεται και αυτή. 121 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική δέλτα υπέρ. Δι. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Αλλά ας κάνουμε μια επαλήθευση. Αφού είναι και συμβαστική. Συμβαστική D λοιπόν. Υπέρ. Ε, μάλλον ε, ε, κλείνω. Εγκρίνεται. Ε υπέρ κατά. Νομίζω θα είναι αναγκαίο να ελέγξουμε. Συμβαστική ε. Κλείνω. Εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. 123 ξανά επαλήθευση. 123. Τέλος. Απερίφθη. 125 υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε και πάλι. 125. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική F. Σίγματα αυτή. Δηλαδή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 και 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική age ή ήτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική α δηλαδή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ. Α, την 134 θέλετε πρώτα επαλήθευση. 134. Εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Εγκρίνεται και αυτή λοιπόν. 136 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε. 142. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική L, λάμδα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική μη, με ονομαστική ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία εδώ. Πέρας. Απερίφθη Υπάρχουν δύο υπέρ. Κατά. Α, μάλιστα εδώ έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία από τους πράσινους. Δύο λοιπόν με ονομαστική. Τέλο Απερίφθη. 13. Υπέρ. Κατά. Προχές. Απορρίπτεται. 12 και 13 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική εν νη υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 14 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται 156 υπέρ, κατά, α, μάλιστα, ας επαληθεύσουμε την 156. 156. Τέλος. Και αυτή απερίφθη λοιπόν. 157. 157, ξαναλέω υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 162 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ κατά ας επαληθεύσουμε. 165 Τέλος. Συμβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R ρο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία τώρα με ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει. Πέρας. Α, μεγάλη υποστήριξη και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα ας προχωρήσουμε στην πρόταση για την εκ νέου χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Εδώ η είναι ο κύριος Σιλικιώτης. Ψηφίζουμε την προσωρινή συμφωνία που έχει επιτευχθεί σε ανεπίσημο τριμερή διάλογο. Ανοίγω την ψηφοφορία, κλείνω την ψηφοφορία. Τεράστια πλειοψηφία, συγχαρητήρια Κύριε Σιγητά, ακολουθεί προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο για Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Μακρόπνο Όραμα για Ευημερούσα Σύγχρονη Ανταγωνιστική και Κλιματικά Ουδέτερη Οικονομία με πολλούς συνεισηγητές. Πρόκειται για τελική ε, ψηφοφορία ονομαστική. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τώρα λίγοι... Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια σε όλους τους συγητές και τις συγγήτριες. Πρόκειται για το ίδιο, προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή. Α, μάλιστα ήταν η προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή. Ωραία. Το ίδιο λοιπόν τώρα για την Επιτροπή. Ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει και τελειώνει τώρα. Σας ευχαριστώ. Μεγάλη υποστήριξη, προφανώς τη βλέπετε. Τώρα, πρόταση ψηφίσματος για το στρατηγικό όραμα κλπ. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο ψηφίσματος αρχίζει. Ονομαστική ψηφοφορία σας τονίζω. Πέρας. Τεράστια υποστήριξη. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρήσαμε θαυμάσια, ομαλότατα έως τώρα. Τώρα, τώρα έχουμε μια γνωμοδότηση. Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας. Εποχικές αλλαγές της ώρας. Σβέν Σούλτσε, ο εισηγητής μας. Να ξεκινήσουμε. 12, 13, 14, 15 από κοινού. Υπέρ. Α, ονομαστική κλίση. Ονομαστική ψηφοφορία λοιπόν. Με συγχωρείτε. Πέρας. Πέρας είπα. Απορρίπτονται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Αγκρίνεται. 6. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. 19 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ, 22, 22, να κάνουμε έλεγχο. Έλεγχο για την 22. Πέρας. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρώτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41-42 υπέρ. Ε, μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά εποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά εποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά εποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά εποχές, απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το ψήφισμα όπως τροποποιήθηκε, τελική ψηφοφορία ονομαστική, πέρας αυτής, εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Και ολοκληρώσαμε με τις ψηφοφορίες για σήμερα. Είναι συνεδρίαση επιτροπής σήμερα το πρωί και το απόγευμα επίσης έχουμε συνεδρίαση. Σας προσκαλώ να έρθετε και το απόγευμα λοιπόν. Now Και τώρα αργά αργά να πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης.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 Ε, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, ας προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, το οποίο είναι okay. Uh, sorry, it's here workshop. E Ομάδα εργασία για την χρήση του υδρογόνου στο μέλλον. Μεταβατική χρήση της ενέργειας στην ε, Γερμανία. Ένα σημαντικό ε, θέμα. Θέλω να καλωσορίσω τους ομιλητές μας. Καθίστε παρακαλώ. Θα ξεκινήσουμε αμέσως. Να καλωσορίσω λοιπόν τους συμμετέχοντες για τη δίκαιη μετάβαση και το παράδειγμα της Γερμανίας επαναλαμβάνω σε τρία τμήματα ο στόχος αυτής της συνάντησης είναι η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που υπάρχουν μέσω της ενεργειακής μετάβασης έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας για να διατηρήσουμε τις θέσεις απασχόλησης. Να εξετάσουμε το ρόλο του υδρογόνου που θα ανοίξει νέες ευκαιρίες στα πλαίσια της ενεργειακής ευελιξίας και διασφάλισης προμήθειας ενέργειας και πώς θα βελτιώσουμε την αποδοτικότητα η οποία θα συνεισφέρει στην απανθρακοποίηση της ε, οικονομίας In general speaking. Okay, great. Λοιπόν, αυτή είναι η στόχη. Έχουμε μία ώρα και 45 λεπτά στη διάθεσή μας για το συγκεκριμένο workshop. 30 λεπτά, ίσως μέχρι 40 λεπτά για κάθε τμήμα. And first session, just energy transition, λοιπόν, το πρώτο κομμάτι της συζήτησης, ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες στα πλαίσια της μεταβατικής περίοδου. Έχουμε τον κύριο Άντρε Φαΐζ, Διευθυντή Σπουδών του μεγαλύτερου οργανωτικού οργανισμού, ε, του μεγαλύτερου ερευνητικού οργανισμού έρευνα ε, των κάτω χωρών. καινοτομίε στον τομέα των ενεργειακών συστημάτων, ε, μέτρα και προτάσεις ε, για τη μείωση της χρήσης του άνθρακα και γενικότερα καινοτομίε στην ενέργεια. Έχουν μεγάλη σημασία τα θέματα αυτά για τη συζήτησή μας. Ο Ολλανδός εκπρόσωπος λοιπόν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε για την εισαγωγή σας. Σας ευχαριστώ όλους που είσαστε εδώ για κάτι το οποίο θεωρούμε και εμείς ότι είναι κεντρικό θέμα τη θέση της βιομηχανίας στην ενεργειακή μετάβαση. Δεν μπορεί να υπάρξει μετάβαση χωρίς την τροποποίηση της λειτουργίας της βιομηχανίας μας είναι ένα μεγάλο κομμάτι των εκπομπών συνολικά, ανάλογα με τη χώρα βέβαια, ποικίλει, αλλά μιλάμε ότι το 1 τρίτο, αν συμπεριλάβουμε και τις έμεσες εκπομπές, ε, οι οποίες ε, χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των ζωοτροφών και η παραγωγή γενικά ενέργειας. Βλέπετε ε, στο γράφημα τις διαφορετικές μορφές ενέργειας οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν εντελώς διαφορετικές διαδικασίες, εντελώς, διαφορετικές, ε, διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας ε, για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και για την παραγωγή ζωοτροφών. Βλέπετε και τεράστια μεγέθη αλλά ταυτόχρονα και τεράστια ποικιλία των τρόπων παραγωγής. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι να βελτιώσουμε φυσικά την ενεργειακή αποδοτικότητα και βλέπουμε εδώ τι δυνατότητες έχουμε στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε ότι σε όλους τους τομείς μπορεί να υπάρξουν βελτιώσεις και στην βιομηχανία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ακραία μέτρα, ήδη έχουν υπάρξει σημαντικές βελτιώσεις προς την κατεύθυνση αυτή στη βιομηχανία αλλά δεν είναι ο μοναδικός τομέας ε, όπου θα βρεθεί η λύση των προβλημάτων. Προσπαθούμε να βρούμε μέτρα πρακτικά όπως η ε, βελτιωμένη άντληση, και βλέπουμε επίσης ε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε τομείς όπως η χαλιβουργία, το τσιμέντο, η αμμονία βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρξουν πιθανές βελτιώσεις γύρω στο 35%. βελτίωση των υπαρχουσών διαδικασιών παραγωγής ή και ε, εφαρμογή νέων. Στη Χαλιβουργία βλέπουμε εδώ ότι ότι υπάρχει η διαδικασία Χισάρνα η οποία χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες μονάδες παραγωγής της εταιρείας ΤΑΤΑ. Βλέπουμε ότι υπάρχει παραγωγή κόκο και υπάρχει μη χρήση των λεγόμενων pellets που χρησιμοποιούνται ε, στη χαλιβουργία παραδοσιακά λόγω ακριβώς της χρήσης ε, του ε, αγνού οξυγόνου μπορεί να υπάρξει παραγωγή χωρίς επιπλέον μόλυνση. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα συλλαμβάνουμε, ε, θα σταματάμε το διοξίδιο του άνθρακα σε μια, βάση, σε μια φάση ε, θα έλεγα πριν από αυτήν ε, την οποία το κάνουμε σήμερα, κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει και την καλύτερη αποθήκευσή του. Τώρα για το CCS οι δυνατότητες και εκεί είναι πολλές έτσι ώστε να μειώσουμε την εκπομπές των παραδοσιακών βιομηχανιών. Εδώ βλέπετε τις εκπομπές ως έχουν σήμερα, ιδιαίτερα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι βασικός στόχος λοιπόν για το CCS. Βλέπετε στο κάτω μέρος του γραφήματος υπάρχει κάτι το καινούριο, είναι το λεγόμενο Bio-Based Conversion ε, και επίσης ε, τα χημικά βιολογικής βάσης. Αυτή τη στιγμή η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τομείς όπως οι υποδομές και οι ζωοτροφές. Είναι μία επιπλέον δυνατότητα για τη μείωση των εκπομπών της βαρέας βιομηχανίας και ιδιαίτερα της χημικής βιομηχανίας. Αν το συνδυάσουμε με την συγκράτηση ποσοτήτων διοξιδίου του άνθρακα, τότε θα έχουμε να κάνουμε με πραγματικά σημαντικότατες αλλαγές. Αυτό φαίνεται επίσης και από άλλα γραφήματα εδώ. Απαιτούνται φυσικά νέες υποδομές για να γίνουν όλα αυτά. Βλέπετε ότι αν έχουμε την λεγόμενη υποδομή CCS θα αλλάξουν τα πράγματα σε σχέση με αυτά τα οποία είναι διαθέσιμα σήμερα το CCS από το μόνο του τα επόμενα 50 χρόνια μπορεί να μας οδηγήσει σε μειώσεις εκπομπών κατά 20%. Ιδιαίτερα στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας όπου υπάρχουν τεράστιες ποσότητες αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα. Τι σημαίνει αυτό τώρα σε κάποια από τα πιο ε, σημαντικά βιομηχανικά κέντρα στο Ράινμοντ, Βλέπετε εδώ λεπτομέρειες πού θα πρέπει να τεθούν οι αγωγοί των αερίων και πώς μπορεί να υπάρξει συνδυασμός των εκπομπών έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε αρκετές πιστώσεις. Η προσπάθεια που γίνεται στην περιοχή Ράινμοντα έχει ακριβώς σαν στόχο την χρήση και την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του CCS. Στα δηληστήρια βλέπετε επίσης ότι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες για να προχωρήσουμε σε μείωση των εκπομπών σε συνδυασμό με το πιθανό κόστος και για την διαδικασία διήλυσης και για τη χρήση της βιομάζας και για τον συνδυασμό με τις μεθόδους ενεργειακής αποδοτικότητας έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μείωση εκπομπών κατά 80% και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να καταλήξουμε σε αρνητικές εκπομπές. Ένα άλλο βασικό θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι η κυκλική οικονομία και εδώ έχουμε την δυνατότητα μείωση των εκπομπών. Έχουμε εδώ τα πρωτογενή υλικά, πρωτογενή ε, στον τομέα της τσιμεντοβιομηχανίας, της βιομηχανίας των πλαστικών κτλ. Οπότε υπάρχει εδώ η δυνατότητα εκμετάλλευσης και ε, ανακύκλωσης ουσιών όπως ε, υλικών συγγνώμη όπως τα πλαστικά, όπως τα τσιμέντα, όλα αυτά βέβαια θα αλλάξουν και τα value chains τα οποία χρησιμοποιούμε στην παραγωγή όπως επίσης και την επιμελητία της μεταφορές και έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε τις ποσότητες πρωτογενών υλικών μέσω ακριβώς της προσπάθειας που θα κάνουμε στην ε, επιμελητιακή αν θέλετε βελτίωση. Έχετε και το θέμα του εξηλεκτρισμού. Βλέπουμε εδώ ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις και σε χημικές διαδικασίες όπως από ε, το ηλεκτρικό ρεύμα στο υδρογόνο, από την παραγωγή ε, ενέργειας στην άμεση παραγωγή θερμότητας, Πολλές φορές ε, απαιτούνται βέβαια συγκεκριμένες καινοτομίες, η χρήση νέων υλικών, καταλυτών και υπάρχουν ε, ανάγκες εδώ για πάρα πολύ σημαντικές καινοτομίες. Αλλά έτσι όμως θα μπορέσουμε να εξηλεκτρήσουμε την βιομηχανία και να καταστήσουμε ταυτόχρονα την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος πιο αποδοτική. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές δυνατότητες εδώ ε, επιλογές όπως σαν παράδειγμα ανανεώσιμες ε, ε, μορφές παραγωγής ζωοτροφών, αποθήκευση επαναλαμβάνω του διοξιδίου του άνθρακα και η έννοια της κυκλικότητας, η ανακύκλωση. Όλα αυτά μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές πάνω από 50%, να φτάσουμε και το 90% το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να βρούμε το, τη σωστή ανάμιξη, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε τον σωστό συνδυασμό, πού θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα CCN εκεί που υπάρχουν, πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος των CCN. Όλα αυτά θα πρέπει να τα αποφασίσουμε την επόμενη δεκαετία. Για να το υπογραμμίσουμε λοιπόν, αυτό από τη μία προσπαθούμε να κάνουμε βελτιώσεις σε επίπεδο μονάδας παραγωγής και να δούμε και πώς αλλάζουν τα δίκτυα της ενέργειας. Εδώ υπάρχουν κάποιοι στόχοι οι οποίοι θα καθορίσουν την εξέλιξη στο μέλλον. Θα ακολουθήσουμε τον στόχο της μείωσης του 95% ή του 80%. Έχουμε διαθέσιμα CCS ή δεν έχουμε. Έχουμε την δυνατότητα ε, χρήσης σταθερής βιομάζας ή δεν έχουμε. Τι γίνεται με το υδρογόνο, τι γίνεται με το υγροποιημένο φυσικό. Όλες αυτές είναι οι επιλογές που θα επηρεάσουν τη μορφή των μελλοντικών συστημάτων. Εδώ βλέπετε ένα διαγράμμα, ε, διάγραμμα ροής που συνδέεται με τις προτάσεις για τη μείωση ενέργειας και χρήσης ηλιακής ενέργειας, αιωλικής ενέργειας. Αυτό θα μπορούσε να είναι το μέλλον. Πάντως αυτή τη στιγμή προωθούμε το CCS που έχουμε διαθέσιμο, προωθούμε τη βιομάζα, το σύστημα αλλάζει και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε, διαφορετικές, σε διαφορετικά κόστη. Βλέπετε ότι τα συστήματα αρνητικών εκπομπών θα μπορούσαν να βοηθήσουν και οι υπόλοιπες, ε, και υπόλοιπους τομείς στην ε, βιομηχανική παραγωγή και το περιβάλλον μέσα στο οποίο τα συστήματα ενέργειας θα πρέπει να αλλάξουν είναι αβέβαια βέβαια και θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες επιλογές. Έχουμε και το σύστημα παραγωγής ενέργειας το οποίο αλλάζει, θα υπάρξουν πιο πολλές διακυμάνσεις λόγω της χρήσης ηλιακής, λόγω της χρήσης αιωλικής και θα πρέπει να υπάρξουν σταθεροποιήσεις σε τομείς όπου θα χρησιμοποιείται υδρογόνο ή θα παράγεται θέρμανση. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε επίσης και χαμηλό κόστος υδρογόνου και αυτό είναι εφικτό αν δούμε ακριβώς τι γίνεται με τη χρήση της ηλιακής και της αιωλικής στο μέλλον τι οικονομίες κλίμακας μπορούμε να κάνουμε, νομίζω ότι θα εξοικονομήσουμε ακριβώς την πράσινη παραγωγή υδρογόνου. Υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις βέβαια για να τα πετύχουμε όλα αυτά και το χρονοδιάγραμμα θα είναι κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό είναι πολύ περίπλοκο το γράφημα αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν διασυνδέσεις και επιρροές ανάμεσα στα εντελώς διαφορετικά συστήματα τα οποία χρησιμοποιεί η βιομηχανία. Αυτές τις αλληλοεπιδράσεις θα πρέπει να τις κατανοήσουμε καλύτερα και έτσι θα πετύχουμε οικονομίες κλίμακα. Έτσι θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε τους τομείς όπου υπάρχει ελκυστική δυνατότητα. Εγώ μιλάω για την Ολλανδία πάντα, στην περιοχή του Δέλτα του Εμς, στο Εμσχάβεν υπάρχουν πάρα πολλές χημικές βιομηχανίες που βασίζονται στην βιομάζα, χρησιμοποιούν επίσης όλο και περισσότερο ε, την εολική ενέργεια από την βόρεια ακτή και υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης επιτόπου της ενέργειας, οι βιομηχανίες τα συνδυάζουν όλα αυτά Υπάρχει λοιπόν ένας τομέας ο οποίος ολοκληρώνεται όλο και πιο γρήγορα στον τομέα της παραγωγής οικολογικής ενέργειας. Ε, προσπαθούμε, υπάρχει και το θέμα του λεγόμενου biorefining ε, που μπορεί να συνδυάσει διαφορετικές πηγές προέλευσης βιομάζας ε, με οικονομικό όφελος. Η δυναμική διαθέσιμη είναι πολύ ενδιαφέρουσα ε, και νομίζω ότι ανοίγει και πάρα πολλές δυνατότητες. Κάποιες τελικές σκέψεις μετά από αυτή την εισαγωγή είναι ότι συνολικά βλέπουμε ότι υπάρχουν επαρκή μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν την απανθρακοποίηση της ε, βιομηχανίας μας και θα μας βοηθήσουν να καταλήξουμε στις αρνητικές εκπομπές. Πολλές από αυτές τις αλλαγές τις οποίες μπορούμε να δούμε σήμερα είναι νέες, είναι καινοτόμες και ακριβώς μπορούν να καταστήσουν τη βιομηχανία μας ανταγωνιστική. Αυτό ε, κατά περίπτωση θα εξετάζεται. Αν το κάνουμε αυτό με τρόπο όχι ιδιαίτερα ευφυή, τότε θα αυξήσουμε το κόστος για τη βιομηχανία και θα μειώσουμε την ανταγωνιστικότητά της. Καινοτομία, ευφυής χρήση των νέων δυνατοτήτων μείωση του κόστους. Κάτι το οποίο θα καταστήσει βιώσιμη οικονομικά την βιομηχανία στο τέλος. Η ανάμιξη των μέτρων αυτών υπόσχεται πολλά. Δεν υπάρχει μία ακραία λύση για όλα τα προβλήματα. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να βρούμε ε, συνδυασμό λύσεων κατά περίπτωση ε, και κυρίως λόγω γεωγραφικής θέσης. Η σταθερότητα ε, της ε, παραγωγής είναι το ζητούμενο. Ε, θα πρέπει να γίνεται σωστή ολοκλήρωση των κύκλων παραγωγής. Θα πρέπει να υπάρχει αξιοπιστία και από πλευράς των ρυθμιστικών αρχών. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους ομιλητές να μην ξεπερνούν τα 10 λεπτά, γιατί τότε δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τις συζητήσεις που θα επιθυμούσαμε. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν. Περνάμε στον επόμενο μιλητή, Μπέμερ, από το Ινστιτούτο του Βούπερταλ. ασχολείστε με συστήματα ενέργειας, ασχολείστε με συστήματα περιβαλλοντικά, και στο Πανεπιστήμιο του Λουν. Εκπομπές ε, ε, αερίου ε, θερμοκηπίων και ουδετερότητα σε επίπεδο επίπτωσης κλιματολογικών αλλαγών και συνεπειών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε καθώς και τους αξιότιμους κυρίες και κύριους ευρωβουλευτές. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσω να συζητήσω μαζί σας για την κλιματική ουδετερότητα, την κυκλική οικονομία, την ενεργειακή μετάβαση, ως ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Δεν θα σας εκπλήξω να δείτε ότι μετά από τους Ολλανδούς έρχονται οι Γερμανοί. Αν δείτε τους χάρτες θα δείτε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κλάστερ ε, στην περιοχή αυτή στο Ρήνο δηλαδή και καθώς ανεβαίνετε προς το βορρά βλέπετε όλο και περισσότερη συγκέντρωση βιομηχανιών εντάσσεως ενέργειας. Όχι μόνο στη Βόρεια Ρενανία Βεσφαλία αλλά σε όλη τη Βόρεια Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία. Είμαστε μια μεγάλη συγκέντρωση λοιπόν τέτοιων βιομηχανιών και αυτό εξηγεί για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ και συζητούμε διεθνώ για τα θέματα αυτά διότι βεβαίως διαβαίνουν τα σύνορα. Θα είδατε και τα σχετικά με το σύστημα CCS και μεγάλες, που, στην Ολλανδία και μεγάλες βιομηχανίες που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακο στη Γερμανία από την άλλη πλευρά, δηλαδή των συνόρων. Άρα το θέμα είναι όντως διεθνές. Εγώ θα επικεντρωθώ σε βασικές βιομηχανίες, basic industries, που είναι πολύ σημαντικές από την άποψη του κλίματος, διότι πέντε βασικά υλικά εκπέμπουν, η, ε, ε, η, η, ε, η παραγωγή τους δηλαδή, χάλιβος, ε, τσιμέντου, πλαστικών, χαρτιού, αλουμινίου είναι υπεύθυνα για παραπάνω από 10 γιγατόνους παγκόσμια. Διοξιδίου του άνθρακος, ε. Στην Ευρώπη η παραγωγή αυτών των υλικών είναι λίγο πολύ σταθερή, όμως παγκοσμίω αυξάνει διαρκώς. Αναμένουμε δηλαδή διπλασιασμό Τη παραγωγής των υλικών αυτών ε, στις επόμενες δεκαετίες. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές σε αυτούς του τομείς. Δεν είναι αδύνατο να γίνει η αποανθρακοποίηση των μεθόδων παραγωγής. Όμω πρέπει να προχωρήσουμε σε πραγματικά ε, δύσκολε ε, λύσει πέρα από την ενεργειακή αποδοτικότητα. και για την άμεση ηλεκτροδότηση και για την έμεση ηλεκτροδότηση. Και βεβαίω ε, αυτό θα είναι και το θέμα του υδρογόνου που θα συζητήσουμε αργότερα. Βεβαίω και την ε, συλλογή και αποθήκευση του, των ε, διοξιδίων του άνθρακο καθώ και την κυκλικότητα τη οικονομία. Πάρα πολύ σημαντικό. Που σημαίνει για να εφαρμοστούν οι στρατηγικέ αυτέ χρειαζόμαστε σημαντικέ τεχνολογίε, σημαντική τεχνολογική πρόοδο πολύ περισσότερο από ό,τι σε άλλου τομεί όπω ε, των οικοδομών, όπου οι βασικέ τεχνολογίε ήδη υπάρχουν. Χρειάζεται λοιπόν να αναπτυχθούν αυτέ οι breakthrough τεχνολογίε και να κάνουμε επενδύσει με υψηλό επενδυτικό κίνδυνο. Αυτό που χρειάζεται βεβαίω είναι και υποδομέ. Όλοι το είδαμε αυτό. Χρειαζόμαστε τεράστιε υποδομέ για τι νέε αυτέ τεχνολογίε που θα χρειαστούν αυτέ οι breakthrough τεχνολογίε και για τη χρήση του υδρογόνου και συστήματα αποθήκευσης του άνθρακο CCS. Και εκεί χρειαζόμαστε επίσης ε, τεράστιες υποδομές. Βέβαια, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις δομές του κόστους, διότι πολλές από αυτές τις μεταποιητικές βιομηχανίες θα αλλάξουν πάρα πολύ βαθιά όταν θα εφαρμόσουμε τις νέες αυτές τεχνολογίες. Θα οδηγήσουν σε μεγάλη αναστάτωση, σε μεγάλες επιχειρήσει. και σε σημαντικές περιφέρειες οι οποίες εξασφαλίζουν μεγάλο όγκο της απασχόλησης. Να έρθω τώρα πάλι στις προκλήσεις. Αν δούμε το χάλιβα, το τσιμέντο και τα χημικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά, οι τρεις αυτοί, αυτοί, τομείς εκπέμπουν 500 εκατομμύρια τόνους ε, του άνθρακο και θα πρέπει να φτάσουν στο μηδέν μέχρι τέλους του αιώνα. Πώς θα γίνει αυτό? Έχουμε σενάρια που σε συνεργασία και με άλλες οδούς, πρώτα-πρώτα την κυκλικότητα και την μείωση της ε, ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε υψηλής ποιότητας χάλιβα με 90% λιγότερη εκπομπή διοξιδίων ε, ε, του άνθρακος. Το ίδιο ισχύει για το αλουμίνιο, όχι όμως για όλα. Και οι προκλήσεις για τα χημικά είναι μεγάλες. Σύμφωνα με τα σενάρια που ακολουθούμε, η κυκλικότητα θα οδηγήσει σε μείωση της τάξης του 20-50% των αναγκών αυτών. Η επόμενη στρατηγική είναι σημαντικό βήμα στην ηλεκτροδότηση. Εκεί πρέπει να ληφθεί υπόψη και το υδρογόνο για τη χαλιβουργία αλλά και για άλλες παραγωγικές διαδικασίες όπως για το τσιμέντο. Και εκεί χρειάζεται σημαντικές αλλαγές στην ανανεώσιμη ε, ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να φτάσουν μεταξύ 44 και 64% της μείωσης των εκπομπών οξυδίων του άνθρακος. Τέλος, η σύλληψη και αποθήκευση του, των οξυδίων του άνθρακος. Εδώ είναι μικρότερη συμβολή αυτής της τεχνολογίας, δηλαδή της τάξης το πολύ μέχρι 25% των συνολικών εκπομπών. Αυτές είναι λίγο πολύ στρατηγικές που έχουμε στα χέρια μας για να μπορέσουμε να αποανθρακοποιήσουμε αυτές τις βιομηχανίες. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε μια συνολική έποψη των βιομηχανιών αυτών, να τις εξετάσουμε από την σκοπιά της κυκλικότητας και από τη σκοπιά των ατομικών συστημάτων ε, καινοτομία, διότι πολλές από τις βιομηχανίες αυτές, για παράδειγμα χημική, η βιομηχανία έχει τη δυνατότητα να ανανεώνεται, αλλά όχι όλες. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες εδώ, αλλά θα προσπαθήσω να σας δώσω μια γεύση του τι σημαίνει η value chain perspective, για παράδειγμα, για το χάλιβα. Όταν μιλούμε για το χάλιβα, μιλούμε για την πρωτογενή παραγωγή του χάλιβα, δευτερογενή ε, ε, ε, του, παραγωγή του χάλιβα και μετά έλαση εν θερμό και εν ψυχρό. Και βλέπετε και τα σχετικά ποσά στον πίνακα. Ξεχνούμε όμως ότι μετά περνούμε στην μεταποίηση, δηλαδή αυτοκίνητα, ε, κατοικίες, κατανάλωση των, ε, των ε, αγαθών αυτών, αποθήκευση πάρα πολλά εκατομμύρια τόνους και βεβαίως ανακύκλωση. Ένα μέρος ανακύκλωσης βέβαια γίνεται αλλού. Έχουμε λοιπόν σε όλη την αλυσίδα αξίας παραγωγή εκπομπών διοξιδίων του άνθρακο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τροχόνο και μπορούμε να μειώσουμε κατά πολύ τι εκπομπέ αυτέ. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και καλύτερα και να ψάξουμε να βρούμε και καλύτερε ευκαιρίε για επιχειρηματικέ ευκαιρίε, δηλαδή για, σε όλε αυτέ τι περιπτώσει, ώστε να ενισχυθεί η αλυσίδα αξιών. Εδώ τέσσερι μπορεί να είναι οι παρεμβάσει. πρωτα Πρώτα-πρώτα στην παροχή ενέργεια, Είναι σαφέ. αν θέλουμε να γίνει από ανθρακοποίηση χρειαζόμαστε πολύ καθαρή ενέργεια. Χρειαζόμαστε πολύ έρευνα και ανάπτυξη και επενδύσει στις νέες τεχνολογίες, πολλέ από τι οποίε ήδη έχουν επινοηθεί, αλλά θα πρέπει να τι φέρουμε σε κλίμακα. Και θα εκεί θα, χρειαστεί πολύ, θα χρειαστούν πολλές επενδύσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορέσει η βιομηχανία να τι χρησιμοποιήσει. Μετά, για να συνεχίσουμε την κυκλικότητα, πρέπει να δημιουργήσουμε την ζήτηση για τα συγκεκριμένα προϊόντα που αρχικά θα είναι πιο ακριβά, πιο δαπανηρά από τα παραδοσιακά. Και τέλος πρέπει να στηρίξουμε την κυκλικότητα, δηλαδή εν τέλει την ανακύκλωση για να κλείσει ο κύκλος στην οικονομία. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα συνολικό πακέτο πολιτικών, βιομηχανικών και κλιματικών πολιτικών που θα ξεκινήσει από το πρώτο βήμα να φτάσει μέχρι το τελευταίο της κυκλικότητας. Αυτού του είδους η καινοτομία λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική χωρίς να λησμονείται και την διαρθωτική πολιτική διότι όλες αυτές οι βιομηχανίες συγκεντρώνονται σε μικρό αριθμό περιφερειών που συνήθως είναι και αυτές που έχουν και τον άνθρακα. Μιλούμε λοιπόν για σημαντικές προκλήσεις και στο περιφερειακό επίπεδο. Και να μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω με έξι συστάσεις, δεν είναι όλες δικές μου, αλλά είναι και από άλλα ιδρύματα του IT50 κλπ. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια εμβληματική αποστολή για προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης για χαμηλό άνθρακα και ούτω καθεξής. Στρατηγική ευθυγράμμιση των βιομηχανιών, των βιομηχανικών μάλλον πολιτικών και ενεργειακών πολιτικών της Ένωσης, της, Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε ε, χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, τα έχω πει αυτά ήδη στην ομιλία μου, για να οδηγηθούμε σε επενδύσεις στις βιομηχανίες αυτές, οι βιομηχανίε αυτέ δεν έχουν επενδύσει πολύ τα τελευταία χρόνια και όπου έχουν επενδύσει το έκαναν περισσότερο στην Ανατολική Ασία και λιγότερο στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε επίση στρατηγικό σχεδιασμό και ανάπτυξη για χαμηλή εκπομπή διοξιδίων του άνθρακο και επομένω για τη σχετική υποδομή. Σχετική, χρειαζόμαστε ρυθμίσει για τη δημιουργία αγοράς και τα προϊόντα των νέων αυτών βιομηχανιών. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας και βεβαίω υπήρξατε και πολύ σύντομο ώστε να μα επιτρέψετε να αρχίσουμε και συζήτηση. Ποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο. Ο κύριος Γκέρεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε, αλλά κάπως ε, μας προκαλέσαν μια σχετική σύγχυση. Θα πρέπει να καθορίσουμε δύο βασικούς προσανατολισμούς ε, από αυτές τις γενικές παρουσιάσεις για να καταλάβουμε προς θα που θέλουμε να πάμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εντοπίσουμε την πραγματική ενεργειακή αποδοτικότητα. Όχι αυτή την οποία αναφέρουν ε, οι κανόνες του κανονισμού. Ήταν λάθος. Λάθος αυτό το, το νομοθετικό εγχείρημα, αυτή η οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα ένα τεράστιο λάθος, διότι δεν έχουμε αποδοτικότητα έτσι, αλλά έλλειψη αυτής. Η αποδοτικότητα, όπως ξέρετε, επιτρέπει τη χρήση της πρωτογενούς ενέργειας που είναι μη ανανεώσιμη, μη ανακυκλώσιμη. Έτσι παράγεται η τελική ενέργεια και έτσι πρέπει να κατανοούμε την αποδοτικότητα. Ε, βάσει της μεθόδου αυτής και του προσανατολισμού μοτοσύσης μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και με βιολογικές ε, μεθόδους, οργανικές. Ε, κάθε χώρα βέβαια πρέπει να κάνει τη δική της την πορεία για να φτάσει προς τα κύρια, αλλά αν αντιπαραθέσουμε την οικονομική αποδοτικότητα των κρατών μελών. Δηλαδή την τελική ενέργεια διαιρεμένη για τις πρωτογενούς προς 100, θα προκύψουν πολλές διαφορετικές συνθήκες. Η Δανία φτάνει στο 80%, η Βουλγαρία ας φτάνει στο 56% με το ζόρι, η Πολωνία είναι περίπου στη μέση, 75% αποδοτικότητας. Άρα θα ήθελα βάσει αυτών των στοιχείων να θέσω και τα ερωτήματά μου προς τους προσκεκλημένους μας. Όχι μόνο με αυτές τις μεθόδους μπορούμε να πετύχουμε την ε, ηλεκτρόλυση, αλλά στα ορυχεία οι δεξαμενές άνθρακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα παραγωγή υδρογόνου με τη χρήση με τη χρήση ε, υδρολογικών πόρων. Αυτή η τεχνολογική λύση δεν είναι η πιο ενδιαφέρουσα όμως αυτή που μας παρουσιάσατε. Θα ήταν ενδιαφέρον εάν ε, χρησιμοποιούσε υδρογόνο. Εντάξει, είδα ότι μου κάνετε νόημα, θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκέρεκ. Αλλά θα θέλαμε, εάν γίνεται ομιλίε και παρεμβάσει να είναι στο δίλεπτο. Διότι έχουμε τρία πάνελ και δεν μπορούμε να πάμε πέρα από τις 12.30. Ο κύριος Έλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις έως τώρα. Υπάρχουν καλά νέα και κακά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι όλα αυτά, δεν υπήρχαν, αυτά που λέτε τώρα δεν υπήρχαν μέσα στις προτάσεις της Κομισιόν για τον ορίζοντα Ευρώπη. Το καλό νέο είναι ότι τα προσέθεσε αυτά στην πρόταση το Κοινοβούλιο μέσω τροπολογιών οι ερωτήσεις που έχουμε κατευθύνονται προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτη, είπατε, σε ό,τι αφορά τη χαλιβουργία, ότι δεν είναι ιδιαίτερα καινοτόμο Από Φάουνχόφερ, Ζαλτσκίτερ και άλλες επιχειρήσεις υπάρχει ένα σχέδιο για την πλήρη τροποποίηση της παραγωγής της ε, χαλιβουργίας Κίτερ με μείωση, σημαντική μείωση των εκπομπών διοξιδίων, των, οξυδίων του άνθρακος κλπ. Και το ίδιο για ολόκληρη την Γερμανία. Υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν σχέδια δηλαδή. Από την άλλη μεριά ο ε, νόμος που ισχύει στη Γερμανία για την τροφοδότηση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος με παραγωγή, παράλληλη παραγωγή, δεν το επιτρέπει. Χρειαζόμαστε λοιπόν project όπου θα κλιμακώσουμε τις προσπάθειες αυτές ή χρειαζόμαστε πραγματικά βασική έρευνα. Τώρα, για τα CCS, μιλήσατε για το ολλανδικό παράδειγμα του CCS. Αν δούμε όμως το δυναμικό που διατυπώσατε, που εξήγησατε κι εσείς, οφείλει να πει κανεί ότι η τεχνολογία δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα χερσαία στην Ευρώπη έχει αποτύχει. Πώς το βλέπετε αυτό τώρα. Πόσο λογικό είναι στην Ευρώπη να υπάρχει μία δομή για την μεταφορά offshore και αποθήκευση των οξυδίων του άνθρακος και κατά πόσο μπορεί να γενικευτεί η προσπάθεια αυτή. Τελευταία παράκληση βρισκόμαστε μέσα στη διαπραγματεύσεις τώρα με το Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικό. Θα μας βοηθούσε πολύ εάν μπορούσατε να απευθυνθείτε και στις ε, κυβερνήσεις των χωρών σας, γιατί βλέπω και η Ολλανδική κυβέρνηση και η Γερμανική κυβέρνηση να είναι πολύ επιφυλακτικές Άρα μην απευθύνετε εκκλήσεις μόνο σε εμάς. Εμείς όλα αυτά τα βάλαμε στα προγράμματα έρευνας. Το ερώτημα είναι θα μπορέσουν τελικώς να συμφωνηθούν ή όχι. Αυτά που προτείναμε εμείς. Ευχαριστούμε κυρία Φανμπρέμπτ. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, αισιόδοξη συμβολή στη συζήτησή μας. Εάν σωστά κατάλαβα όπω είπατε, υπάρχουν ακόμα κάποιες αμφιβολίες για το ποιο θα πρέπει να είναι η σωστή ανάμειξη, το μείγμα το ενεργειακό των διάφορων λύσεων. Αυτά είναι καλά νέα βέβαια ότι μπορεί να έχουμε κάποιο χρόνο μπροστά μας για να προσαρμοστεί η βιομηχανία. Αλλά μερικές πρακτικές ερωτήσεις ίσως το 2030 και 2050 αφού έχουμε κάποιο χρονικό περιθώριο. Ως πολιτική Πρέπει να ξέρουμε τι ρυθμιστικό πλαίσιο ε, πρέπει να δημιουργήσουμε. Εγώ είμαι από την Αμβέρσα και υπάρχουν ε, προγράμματα για ένα νέο χημικό εργοστάσιο στην Αμβέρσα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε εάν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες ταιριάζουν με αυτά που μας λέτε. Εάν χρησιμοποιήσουμε, αν χτίσουμε μάλλον ένα χημικό εργοστάσιο με τη σημερινή τεχνολογία, πόσο αποδοτικότερο θα είναι το πρόγραμμα αυτό ε, βάσει των όσων προσφέρονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και σε σχέση με τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε μελλοντικά. Σε ό,τι αφορά το CCS και το CCU, θα πρέπει μάλλον να επιβάλλουμε αυτή την τεχνολογική λύση ως προϋπόθεση για το χτίσμα αυτών των εργοστασίων. Είναι πολύ ακριβή και δαπανηρή η επιλογή. Χρησιμοποιείται αλλού στην Ευρώπη αυτή η ερώτησή μου. Διότι θα χρειαστεί να ε, πιεστούμε για να την εφαρμόσουμε. Και πώς γίνεται όλοι να πληρώσουν ένα ακριβό ποσό εκ των προτέρων για να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια τεχνολογική λύση. Ας πούμε, σε αυτή τη θητεία του Κοινοβουλίου εγκρίναμε και το σύστημα ανταλλαγή δικαιωμάτων εκπομπών, αλλά Α σκεφτούμε και τη φορολόγηση γενικότερα. Πρέπει να προβλέπουμε και άλλους φόρους, φόρους διεξουδίου του άνθρακα, διότι τότε θα βρούμε τα κατάλληλα κονδύλια, του σπόρου που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε σε αυτέ τι επενδύσει. Ευχαριστούμε ο κύριο Γιάβορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ και του ομιλητέ που μα ανέπτυξαν τι απόψει του για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Έχω μία ερώτηση. Μία ερώτηση που όλοι σα, ε, καθώ μιλήσατε, την αναπτύξατε. Είπατε για ένα διαφορετικό ενεργειακό μείγμα των διάφορων τεχνολογικών λύσεων στην ουσία. Το CCS, το CCU, το υδρογόνο και την κυκλικότητα. Όμως η πραγματική ερώτηση από την πλευρά τη αγοράς είναι ποιο είναι το κόστος των διαφορετικών επιλογών. Αντί να προσπαθούμε να προτείνουμε διαφορετικά μείγματα, ίσως ως νομοθέτε, πρώτα πρέπει να δούμε ποιο είναι το κόστος των διαφορετικών τεχνολογικών λύσεων και πώς μπορούμε να μειώσουμε αποτελεσματικά τις εκπομπές της βιομηχανίας μας. Πηγαίνοντας δηλαδή προς την κυκλική οικονομία, ε, είναι καλή ιδέα να πάμε προς το CCG και το CCS, γιατί για την ώρα είναι πολύ ακριβή τεχνολογία. Πείτε μας λοιπόν το κόστος των διαφορετικών τεχνολογικών λύσεων και πώς θα μπορούσαν όλα αυτά να ενταχθούν στις ανάγκες της βιομηχανίας μας με ενόψη της κυκλικότητας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Ο κύριος Κλέτς, για το θέμα της κυκλικής οικονομίας. Είπατε και οι δύο ότι είναι σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομία ως το 2050 να υπάρξει σωστή μετάβαση. Πρέπει όμως να έχουμε κάποια νομοθεσία για τα αστικά απόβλητα. Τα αστικά λύματα μάλλον. Εκεί Μπορεί να χρειαστούν και νέε υποδομες υποδομές. κάτι κράτη-μέλη προχωρούν στην αποτέφρωση για την ε, αποκομιδή των αστικών λιμάτων, ενώ κάποιοι προχωρούν στην, ε, στην ε, πανεπεξεργασία ή ταφή. Εδώ λοιπόν για τα βιομηχανικά απόβλητα, στην περίπτωση του αλουμινίου, του σιδήρου, Τη σχετική βιομηχανία και των εξαγωγών της εκτό Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πιο κερδοφόρο για τις εταιρείε που έχουν τέτοιου είδου απόβλητα να πουλάνε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή οι δυνατότητέ μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ξεπερασμένε. Ε, δεν χρησιμοποιούνται επαρκώ. Και επίση είναι ένα θέμα και η νέα τεχνολογία που αναφέρατε. Οι καινοτομίε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι υπάρχει μια, εδώ μια αντιπαλότητα μεταξύ του δημοσίου συμφέροντο. διότι είμαστε μεν υπέρ τη συμφωνία των Παρισίων να μειώσουμε τι εκπομπέ του θερμοκηπίου, αλλά, των αερίων του θερμοκηπίου, αλλά χρειαζόμαστε και αυτέ τι νέε τεχνολογικέ λύσει. Θέλουμε να είναι προσιτέ όμω. Και όχι μόνο στο πλέον ανεπτυγμένο μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για όλου. Διότι το πρόβλημα τη τεχνολογική λύση στον τομέα των ανανεώσιμων είναι ότι είναι φθηνέ και προσιτέ μόνο στου πιο πλούσιου τη Ευρώπη, όχι στου υπόλοιπου. Και το δεύτερο είναι για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων. Μιλήσατε για τα προβλήματα της τσιμεντοβιομηχανίας και άλλων κλάδων που έχουν να κάνουν ακριβώ με τα μεγάλα κτίρια στις δικές σας ε, τις εκτιμήσεις, πώς βλέπετε την αλλαγή των ε, υλικών που χρησιμοποιούνται για τα κτίρια. Θα έπρεπε να χρησιμοποιείτε ξύλο αντί για τσιμέντο ή τούμπαλιν. Και όχι μόνο σίδερος και τσιμέντο. Ε, πρέπει δηλαδή να αντικατασταθούν οι πρακτικές μας. Επίσης, μεταφορές είναι ένα άλλο θέμα. Σήμερα διάβασα ότι η Ουγγαρία έκλεισε μια συμφωνία για τα φορτηγά. Καλά, καλά, θα ολοκληρώσω. Πώ βλέπετε και αυτό το κομμάτι. Και τέλο. ποιο είναι το πρόγραμμα που βλέπετε. Ε, ποιο χρονοδιάγραμμα βλέπετε για τα σενάρια που αναπτύξατε, Ποιο είναι αυτό που πρέπει να προτιμούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ, φίλοι μου, αλλά έχουμε τέσσερι ακόμα ομιλητέ μετά. Μην το ξεχνάτε. Ακούσαμε όλους τους ε, ομιλητές που είχαν ερωτήσεις για το πρώτο πάνελ. Παρακαλώ να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ για τις εξαιρετικές ερωτήσεις σας. Καλό θα ήταν να μπορούσα να απαντούσα ε, αναλυτικά σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά δεν είναι δυνατόν να το κάνω. Καταρχάς χαίρομαι γιατί βλέπω ότι κατανοείτε την περιπλοκότητα της κατάστασης και πώς συνδέεται με την καθημερινή πολιτική και τις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων σε τομείς όπου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με τέτοια θέματα περισσότερο από ό,τι και στις ισχύουσες οδηγίες. Αυτό θα μας επιτρέψει στο να μετακινήσουμε τις πολιτικές μας και να πετύχουμε μειώσεις ε, ε, στις εκπομπές συνολικά και όχι μόνο στην μείωση, ε, στην mm. προσπάθεια επίτευξης συγκεκριμένων επιμέρους στόχων. Είναι καλό να υπάρξει μια συνολικότερη, αν θέλετε, αντίληψη για τα πράγματα. Αν το πετύχουμε αυτό, τότε θα mm. ξεκινήσουμε να βλέπουμε και κάποιες απαντήσεις σε επίπεδο μονάδας παραγωγής, σε επίπεδο περιφέρειας, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές λύσεις, αναλόγως με τις ευκαιρίες. Το CCF δεν είναι παρόν πάντα. Η διαθεσιμότητα βιομάζας είναι καλή σε ορισμένους τομείς, σε άλλους τομείς, σε άλλες περιφέρειες δεν είναι και γι' αυτό ακριβώς οι υπολογισμοί μας δείχνουν συστηματικά θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι κανείς πραγματιστής και δει τα πράγματα μακροπρόθεσμα και δει ποιοι είναι οι στόχοι μακροπρόθεσμα, τότε μπορεί να πάρει κάποια βήματα και εύραχη πρόθεσμα. Κάποια μπορεί να γίνουν στην παρούσα φάση, κάποια πρέπει να καθυστερήσουν γιατί πρέπει να είναι διαθέσιμη η τεχνολογία. Αυτή η ευελιξία είναι κάτι το απαραίτητο έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε με σωστό τρόπο τα πλαίσια στα οποία κινούμεθα και συμφωνούμε πλήρως ότι η καινοτομία στην βιομηχανία και η καινοτομία στις υποδομές της ενέργειας είναι βασικές. Είμαστε σε διαδικασία μαθητείας για τις μεθόδους μείωσης του κόστους. Έχουμε πολύ καλά επιτεύγματα στον τομέα της μείωσης του κόστους στην ηλιακή και στην αιωλική και μπορούμε να επαναλάβουμε τα κόλπα αυτά αν θέλετε, τα μαθήματα αυτά και για το CCS και για την βιομάζα και υπάρχει μια κατανομία, κα, κατανόηση ανάμεσα στη βιομηχανία και την ενέργεια στην Ευρώπη. Αυτό όμως προϋποθέτει σταθερότητα και σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο καινοτομίας. Νομίζω ότι έχουμε κάποια καλά παραδείγματα των συνεργασιών που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που στηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας αφήσουμε ας πούμε ε, τις βιομηχανίες του Χάλιβα να συνεργαστούν σωστά, τις βιομηχανίες φυσικού αερίου να δουλέψουν καλύτερα για τους ηλεκτρολίτες και να τους καταστήσουν ευθυνότερους. Όλα αυτά ε, είναι πράγματα τα οποία θα, ε, θα πιέσουν προς τη σωστή κατεύθυνση και θα δούμε πώς αυτές οι επιχειρηματικές επιμέρους περιπτώσεις συνολικά θα προσθεθούν και θα βοηθήσουν ακριβώς να προχωρήσουμε. Ε, έχουμε λοιπόν την δυνατότητα σήμερα να βελτιώσουμε τις καταστάσεις, τις διαδικασίες ε, συγκράτησης του διοξιδίου του άνθρακα. Ε, το κόστος αυτής της συγκράτησης είναι ιδιαίτερα υψηλό με τις διαθέσιμες και τεχνολογίες ε, θέλουμε να βελτιώσουμε λοιπόν την κατάσταση αυτή τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον κατά 10%. Αυτό με τον σωστό προγραμματισμό και οι υποδομές εδώ παίζουν ρόλο και εδώ απαιτείται καλύτερο συντονισμός ανάμεσα στις κυβερνήσεις και οι περιφερειακές συνεργασίες και η ανάπτυξη των δικτύων υποδομών ως έχουν σήμερα ε, σε πολυμερή βάση, σαν παράδειγμα στη Βόρεια Θάλασσα, ξέρουμε ότι θα υπάρξει εξοικονόμηση πιστώσεων αν υπάρξει συντονισμένος τρόπος αντιμετώπισης. Ή ε, ιδιαίτερα και στα προβλεπόμενα σχέδια για παραγωγή ολικής ενέργειας που θα φτάνει τα 2,5 ε, γιγαβάτ. Αυτό θα εξοικονομήσει μακροπρόθεσμα πάνω από 2,5 δις Συνεπώς λοιπόν απαιτείται να συνεργαστούμε για να πετύχουμε τους στόχους. Προς το παρόν λοιπόν έχουμε την συγκεκριμένη προοπτική. Ας αφήσουμε τη βιομηχανία να παίξει τον ρόλο της, ας αφήσουμε τις επιμέρους περιπτώσεις να αναπτυχθούν, ας μην ξεχάσουμε ότι η βιομηχανία η χημική στην Ευρώπη είναι από τις ισχυρότερες στον κόσμο. Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία, εξαιρετικά προοδευμένες χημικές ε, βιομηχανίες. Είναι αβέβαιος όμως ε, οι εξελίξεις γιατί δεν έχουμε ευθυνό αέριο, δεν έχουμε ευθυνό πετρέλαιο, ε, αντίστοιχες φθηνές παραγωγές παραδοσιακής ενέργειας υπάρχουν στην Ανατολική Ασία, υπάρχουν στην Βόρεια Αμερική και θα πρέπει να αντικαταστήσουμε αυτή την διαθεσιμότητα που είχαμε μέχρι σήμερα έτσι ώστε να είμαστε παρόντες σε ηγετική θέση ε, και στο μέλλον. Αυτό είναι αν θέλετε σε οραματικό στάδιο στόχος. Ακούω πολλές βιομηχανίες οι οποίες θέλουν όμως να δουλέψουν προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν τις καινοτομικές δυνατότητες, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούν με, τις, ε, ε, με τα δίκτυα, τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας, λέει ο κύριος Λεχτενμπέμερ. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος η Ευρώπη να μειώσει αυτή τη δραστηριότητα στο μέλλον, πιέζεται η Ευρώπη και ακριβώς η πρόοδος προς την κυκλική οικονομία και την μείωση της χρήσης του άνθρακα είναι κάτι το οποίο ανοίγει ευκαιρίες. Ίσως να είναι η τελευταία ευκαιρία. Τώρα απαιτείται φυσικά η καινοτομία σε όλους τους τομείς και στην κυκλικότητα και στις νέες, ε, ε, στους νέους τομείς. Απαιτείται όμως και κλιμάκωση ε, των ενεργειών, απαιτούνται επιστώσεις στην πρώτη φάση και εδώ η μόχλευση από πλευρά της Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικότατη για την καινοτομία και θα πρέπει να ε, βοηθήσουμε τις επενδύσεις στον τομέα. Απαιτούνται, ε, ε, θα έλεγα, σημαντικότατες επενδύσεις για να προωθηθεί η βιομηχανία αυτή. Ένα άλλο θέμα είναι η χρήση του υδρογόνου στην χαλιβουργία. Οι χαλιβουργοί έχουν πει ότι θέλουν να ακολουθήσουν την πορεία αυτή εγώ δεν έμεινα στο σουηδικό παράδειγμα, αλλά περιμένουν ότι θα μπορούσε να υπάρξει δυνατότητα παραγωγής και χρήσης του υδρογόνου μάλλον με κόστος μόνο 20%, κάτι το οποίο με άλλες εξοικονομήσεις κλίμακας θα κρατούσε το σουηδικό χάλιβα σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Συνεπώς λοιπόν αυτά δεν πρέπει να μείνουν στα χαρτιά όπως είναι τώρα, το θέμα είναι να προχωρήσουν οι βιομηχανίες και αυτό θα εξαρτηθεί από τις διαθέσιμες υποδομές. Αυτό το οποίο χρειάζονται οι επιχειρήσεις είναι υψηλές ποσότητες πράσινου υδρογόνου και εδώ έχουμε ανάγκη από άλλες τεχνολογίες για την παραγωγή του πράσινου υδρογόνου. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες αυτές. Τώρα για την συγκράτηση του διοξιδίου του άνθρακα και την αποθήκευση. Εξαρτάται που βρίσκεται κανείς. Οι προτάσεις μου αποτελούν μια κατελάχιστον λύση. Ας πούμε η, τσίμπενο, η τσίμεντοβιομηχανία μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να συνδράμει. Η βιομάζα, εκεί ίσως είναι μικρότερες οι δυνατότητες. Υπάρχει όμως η δυνατότητα του CCS τα έχουμε συζητήσει αυτά στο παρελθόν και για την ηλεκτρική ενέργεια. Το CCS και το CCU είναι ήδη τμήμα της λύσης, αλλά θα πρέπει να είναι οι λύσεις αυτές προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες. Και για τα κόστη τώρα. Προφανώς όλα αυτά κοστίζουν πάρα πολύ και δεν είναι εύκολο να αποφασίσει κανείς ποιος είναι ο σωστός δρόμος Νομίζω ότι απαιτούνται πολιτικές αποφάσεις έτσι ώστε να δούμε πώς πηγαίνουν οι αγορές οι οποίες δεν μπορεί να είναι τόσο ταχύες όσο επιθυμούσαμε. Το πλαστικό μπουκάλι, ένα πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιείται από άνθρακα από το CCU και από ανανεώσιμη θα έλεγα πηγή ενέργειας έχει διπλό κόστος. Αυτό θα διώξει τον κόσμο από την αγορά. Από την άλλη βέβαια το κόστος αύξησης του τελικού προϊόντος θα είναι ελάχιστο ε, σε ένα μπουκάλι σαμπουάν ας πούμε. Ε, λοιπόν, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε για να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις αυτές της αγοράς, πώς μπορούμε να καινοτομήσουμε. Δεν έχουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα, ακόμα και σε επίπεδο διανοητικών ε, προτάσεων αν θέλετε. Νομίζω ότι ε, καλό θα είναι να πληρώσουμε κάτι παραπάνω για ένα μπουκάλι σαμπουάν έτσι ώστε να αποφύγουμε τα προβλήματα που δημιουργεί η παραδοσιακή παραγωγή πλαστικών μπουκαλιών. Σας ευχαριστώ για τις εξαιρετικές σας παρεμβάσεις και εγώ είχα τρεις-τέσσερις ερωτήσεις αλλά παρετήθηκα γιατί θα πρέπει και οι υπόλοιποι να πάρουν το λόγο. Σας ευχαριστώ όλους. Μόλις τώρα ξεκινάει η συζήτηση αυτή, βρισκόμαστε στην αρχή. Έχουμε δύο ομιλητές ακόμα. Ο ρόλος του υδρογόνου στο μέλλον. Ο κύριος Πολ Τότς είναι ο πρώτος από το UCL στο Λονδίνο και ο πρώην Ευρωβουλευτής και τη επίτροπή Ήτρε, ο κύριος Γιώργο Χατζημαρχάκης. Δεν χρειάζεται να σας συστήσουμε καν στα μέλη τη Επιτροπή. Ας περάσουμε ευθύ αμέσω στην πρώτη ομιλία και λόγο τον κύριο Πολ Τότζ να ακούσουμε, τον καθηγητή, δόκτορα, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερως με τη χρήση και τον εξυγχρονισμό των διαφόρων ε, συστημάτων ε, με υδρογόνο την ενεργειακή αποθήκευση, το σχεδιασμό ενεργειακών μοντέλων που βασίζονται στο υδρογόνο, το μέλλον των δικτύων ε, φυσικού αερίου του Ηνωμένου Βασιλείου, την μετάβαση σε μια οικονομία που καταναλώνει λίγο άνθρακα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τα θέματα ασφάλειας στην πυρηνική βιομηχανία. Πάρα πολύ ευρέα τα θέματά σας, αλλά εδώ μας ενδιαφέρει το μέλλον τη στο, ο ρόλος του υδρογόνου στο μέλλον. Ευχαριστώ. Όπως καταλάβατε είμαι λίγο πολύ, ασχολούμαι με όλα εδώ. Και σας ευχαριστώ πολύ για την ε, ωραία αυτή σύσταση αλλά βλέπετε τον τίτλο του ομιλίας, ο ρόλος του υδρογόνου στο μέλλον. Ασχολούμαστε με όλες τις διαστάσεις του υδρογόνου, την αποθήκευση, την ε, χρήση του, τη διαδικτύωση και το καθεξής. Αυτά σας τα λέω γιατί νομίζω ότι πραγματικά έχω μια ευρεία ε, έποψη του ενεργικού συστήματος και το στόχος είναι πώς μπορεί το υδρογόνο να ενταχθεί σε όλο αυτό το σύστημα. Γι' αυτό φτιάχνουμε και τέτοιου είδου μοντέλ ενεργειακά συστήματα. Πολλοί τα βλέπουν σαν κουτάκια, φανταστείτε και το γιατί, αλλά ο στόχο είναι πώ να απαλλάξουμε την οικονομία από τον άνθρακα με το χαμηλότερο δυνατό κόστο. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τι μα λένε αυτά τα διαγράμματα. Εδώ είναι ένα τεχνολογικό σενάριο με 80% μείωση στη στέρεο θερμοκηπίου και το Ηνωμένο Βασίλειο και το παράδειγμα που προκύπτει. Να ένας τρόπος να απαλλαγεί από τον ανθρακά Βασίλειο. Βρήκαμε ότι το 2050 μπορούμε να έχουμε 24% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας λιγότερο, χάρη στο υδρογόνο. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι 40% για τη βιομηχανία. Και μετά υπάρχουν άλλα δύο μεγάλα κομμάτια για τη θέρμανση, ε, για τον κλιματισμό στον τομέα της στέγασης και τις μεταφορέ αλλά έχουμε 400 πετατζά ολυδρογόνους σε αυτή την περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Και εδώ έχουμε ένα σενάριο από δημοσίευση τη Times και των φίλων μου του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου. Βρήκαν ότι για τις μεταφορές μπορεί να έχουμε μια ε, μείωση με 500 πετατζά ολυδρογόνου στις μεταφορές. Ωραίο και για το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούσε να γίνει αλλά πρέπει να γίνει κάτι ε, και για την ε, θέρμανση των κτηρίων που δεν υπάρχουν ακόμα στα μοντέλα. Να, εδώ λέμε για τα καύσιμα των αυτοκινήτων και τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα. Είναι η κυρία για το υδρογόνο στα καύσιμα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να πάει κανείς ένα ε, όχημα που να κινείται με υδρογόνο. Να αυτό το καύσιμό του είναι κάτι που έχει αρχίσει πολύ τα δύο τελευταία χρόνια. Τώρα η μεγάλη κλίμακα παραγωγή ε, στην Αποανατολή έχει προχωρήσει με την τελευταία διετία μόνο. Και όταν λέω μεγάλη κλίμακα, εννοώ χιλιάδε αυτοκίνητα συνέχεια. Αλλά υπάρχουν και άλλε αγορέ που αρχίζουν να ανοίγουν για τα οχήματα που χρησιμοποιούν υδρογόνο, τα ε, lift, αυτά που κάνουν μεταφορέ, τα φορτηγά, τα ελεφορία και τα τρένα στη Γερμανία ιδίω. Στο μοντέλο μα δεν είχαμε Πολλέ υδρογονικές μεταφορές. Σε πολλά από τα σενάρια που είδαμε από διεθνεί οργανισμού και φορείς ή την Επιτροπή των Κλιματικών Αλλαγών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είδαμε ότι η ενεργειακή βασιλειο ειδαμε οτι η ραγικη μεταβαση θα ε, κυριαρχήσει στην αγορά, αλλά ήδη έχει κυριαρχήσει στην αγορά και θα αλλάξει κι άλλο. Τώρα, για το KPMG που είναι ε, ε για τα αυτοκίνητα για την αυτοκίνηση και για την έρευνα που παρήγγειλε το 2019, μελέτησε τα ηλεκτρικά οχήματα. Είδε ότι είναι 71% θα έχει συμφωνηθεί σε 71% χρήση στην Ευρώπη. Και όσο πιο ε, ψηλά βρίσκεται κανείς ε, την, ε, στην εταιρεία αυτή που ασχολείται με, τα, με την αυτοκίνηση, την κίνηση δηλαδή με την κυκλοφορία με αυτοκίνητα έχει και διαφορετικές απαντήσεις. Τώρα, το Συμβούλιο του Ιδρογόνου έχει πολλά ενθουσιώδη μέλη. Είναι πολύ αισιόδοξοι αυτοί που συμμετέχουν εκεί. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική επιστημονική, ε, δεν υπάρχουν εναλλακτικά επιστημονικά στοιχεία για το πόσο το υδρογόνο θα μπορεί όντω να αντικαταστήσει τα ηλεκτροκίνητα οχήματα στο μέλλον. Εδώ μια μικρή παρουσίαση για το τι θα είναι ένα, με τι θα μοιάζει ένα αυτοκίνητο που θα κινείται με καύσιμα και τη διαφορά με τα, υδρογόνου, τα κινούμενα με υδρογόνο και τα, αυτά που κινούνται με μπαταρίες. Ε, η μπαταρία αντικαθιστά τη δεξαμενή του καυσίμου. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές δυνατότητες σχεδιασμού. Ε, για τα υβριδικά, απλώς η διαφορά θα είναι η δεξαμενή υδρογόνου σε σχέση με αυτά που έχουν την... Ε, Όλα έχουν όμως μπαταρία. Βλέπουμε ότι το κόστος είναι κάτι που δεν ε, μπορεί να καλύψει το διάγραμμα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι το πάνω μέρος ε, του της στήλη είναι τα καύσιμα, το κόστος του καυσίμου. Είναι πολύ μικρό το κόστος της συνολική τιμής που έχει να κάνει με τα υπόλοιπα. Το δυσκολότερο είναι να πληρώσει κανείς το αρχικό κόστος ε, για το καύσιμο και μετά για να συντηρεί και να κινεί το όχημα. Αυτό είναι το πιο ακριβό κομμάτι. Εάν κοιτάξουμε τώρα το κόστος της παραγωγής αυτών των ε, οχημάτων, το διάγραμμα μπορούμε να το δούμε ως προς το συνολικό κόστος κατοχής από αυτό το πρίσμα. Και εδώ έχουμε κάποιε προβλέψει για το πώ θα μπορούσαν να δημορφωθούν τα πράγματα. Είναι λίγο αβέβαιο για το, το τι θα γίνει με το κόστο τεραγών στο μέλλον, αλλά αυτό που βρίσκουμε είναι ότι ε, από το 2030 και μετά όλες οι δυνατότητες ε, ενεργειακών ε, μάτων που αναφέρονται στο παρελθόν θα έχουν ένα μεγάλο κόστο. Και πρέπει να αποδεχτούμε ότι το κόστο πολλών από αυτέ τι τεχνολογικέ λύσει είναι αβέβαιο. Αλλά επειδή το κόστο είναι τόσο ασταθέ, αυτό που προκύπτει από το διάγραμμα είναι ότι δεν ξέρουμε καθόλου ποιε θα είναι οι φθηνότερε τεχνολογικέ λύσει στο μέλλον. Δεν έχουμε ιδέα. Αλλά αν το κόστο συγκλίνει κατά αυτόν τον τρόπο, το θέμα της προσφοράς οχημάτων, του χρόνου ε, τη γεμίσματος της δεξαμενής, το κατά πόσον θα υπάρχει έλλειψη χώρου στα σπίτια. Αυτά θα είναι θέματα που δεν έχουν να κάνουν το κόστος και θα γίνουν πολύ πιο σημαντικά. Είναι πολλοί αυτοί που θα πληρώνουν κάτι παραπάνω για να... Ε, καταφέρουν ε, κάτι από όλα αυτά. Δεν είναι δύσκολο λοιπόν να κάνουμε τώρα τη σωστή επιλογή όταν δεν ξέρουμε ποια θα είναι η καλύτερη λύση στο μέλλον. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο διάγραμμα που δείχνει καινοτομία στο, στη θέρμανση και την πώληση των ε, μπαταριών στην Κορέα και την Ιαπωνία. Βλέπουμε ότι όσο αυξάνεται η πώληση πέφτει η τιμή. Άρα η καινοτομία δίνει αποτελέσματα. Δεν το έχουν καταλάβει περισσότερο με τις, με τις μπαταριών δεν έχουν καταλάβει ότι οι μπαταρίε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη θέρμανση και όχι μόνο για την Ευρώπη. Πού βρίσκεται λοιπόν η Ευρώπη μέσα σε όλα αυτά. Εδώ βλέπουμε τι γίνεται με τα διπλώματα βρεσιτεχνία. Ε, όχι με τη χρήση του. Ε, σε πολλέ χώρε το πρώτο που μπορεί να προσέξει κανεί είναι η διαφορά μεταξύ των δύο διαγραμμάτων. Πάνω έχουμε τα ρεκτά καύσιμα. Μετά βλέπουμε την χρήση του υδρογόνου στι μπαταρίε για τι μεταφορέ. Εδώ είναι πιο σημαντικό. Και βλέπουμε ότι ο αριθμό των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία μειώνεται. Διεθνώ. Ενώ η χρήση του αυξάνεται. Το δεύτερο που μπορούμε να αποδεχτούμε είναι ότι η Ιαπωνία και η Κορέα έχουν πολύ περισσότερα διπλώματα βιοτεχνία από ό,τι ευρωπαϊκέ χώρε. Η Ευρώπη δεν είναι σε πρωταγωνιστική θέση. Δεν είναι πρωτοπόρο. Επίση, πρέπει να σκεφτούμε την κυβερνητική στήριξη και το πώ αναπτύσσονται αυτέ τι λύσει συνολικά. Παίρνω ένα παράδειγμα, την Ενωμένη Βασιλεία και τη Γερμανία. Βλέπουμε ότι η Ιαπωνία έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για τη χρηματοδότηση. Για τη θέρμανση των οχημάτων και τα οχήματα. Στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε κάποια προσπάθεια, αλλά δεν πλησιάζουν καν κοντά στην Ιαπωνία. Έχουμε μείνει πίσω. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Our next speaker, uh, ναι, σπιτιών. Um, Ευχαριστώ λοιπόν. Τώρα μετά από τις θητείε του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Γιώργο Χατζημαρκάκη είναι μαζί μα. είναι Γενικός Γραμματέας της Hydrogen Europe από το 2016 και χάρη στην μεγάλη σου εμπειρία συνέβαλες για να μπουν τα θεμέλια του πρώτου και δεύτερου κοινού undertaking για τη χρήση του υδρογόνου. Αυτά τα joint undertakings, οι ε, συνεργασίες, οι κοινοπραξίες δηλαδή, ε, ήδη αναφέρθηκαν τους προηγουμένους ομιλητές. Γιώργο, έχεις τον λόγο και θα ομιλήσεις για το υδρογόνο στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Ζέρζη. Βέβαια, είναι πράγματι συναρπαστικές οι εξελίξεις στον τομέα αυτό, όπως εξήγησε και ο καθηγητής Dodge πολλές επιχειρήσεις, θα σας τις δείξω τώρα. Εμείς είμαστε μέρος όλης αυτής της υπόθεσης που βλέπετε εδώ. Το λέω στους ευρωβουλευτές ότι υπάρχει και μια δεύτερη ζωή. Η γυναίκα μου κατεβαίνει υποψήφια για ευρωβουλευτής, άρα η οικογένεια θα συνεχίσει να είναι. Ε, εγώ όχι. Αυτό το, αυτή η κοινοπραξία που βλέπετε εδώ είναι μια κοινοπραξία, αν θέλετε, μεταξύ του δημόσιου τομέα, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εκπροσωπείται εδώ, στην ε, παρούσα αίθουσα. Βλέπω δηλαδή με χαρά μου ε, εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και από την άλλη μεριά της βιομηχανίας και της έρευνας. Έχουμε πολλά επιτυχή project ε, για τη μεταφορά ενέργειας, αλλά και οριζοντίω. Ποιο είναι ο ρόλος του υδρογόνου. Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό να κατανοήσει κανεί τους 7 διαφορετικούς ρόλους του υδρογόνου. Και γιατί είναι τόσο μεγάλο το θέμα του υδρογόνου. Δεν πρόκειται για τεχνητή ε, αύξηση ή τεχνη, τεχνητό τονισμό του ρόλου του, αυτό το hype. Το ε, υδρογόνο έρχεται και θα μείνει είχαμε πριν από μια εβδομάδα στο Παρίσι ότι και μας είπαν το υδρογόνο έρχεται και θα μείνει. Ο το πρώτος του ρόλος είναι να επιτρέψει σε μεγάλη κλίμακα την ένταξη των ανανοσίμων πηγών ενέργειας στα συστήματα παραγωγής ενέργειας. Εδώ περισσότερες ανανεώσιμες χρειάζονται και περισσότερο χώρο αποθήκευσης. Δεύτερο, η διανομή οριζοντίως μεταξύ τομέων αλλά και μεταξύ περιφερειών. Για τους τομείς θα σας τα πω, αλλά για τις περιφέρειες είναι απλό. Αν μεταφέρετε ένα ηλεκτρόνιο που έχει, που έχει ε, παραχθεί ε, είναι 20 φορές 100 περισσότερο από το να μεταφέρει σε ένα ε, μόριο αερίου. Άρα λοιπόν είναι το ζήτημα να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς. Και από την άλλη μεριά είναι και μια ζώνη προστασίας ανάμεσα στην παραγωγή και στο σύστημα διανομής. Άρα αυξάνει την ανθεκτικότητά του. Μπορεί μετά να αποανθρακοποιήσει και τους τελικούς χρήστες. Αφενός στις μεταφορές, αλλά και στην βιομηχανική χρήση της ενέργειας, ε, στη θερμάνση οικοδομών κλπ. Και τέλος, το υδρογόνο ως ζωοτροφή. Αυτά με συγχωρείτε, ως φίτστο όχι ζωοτροφή, αλλά ως, ε, για τη χρήση μάλλον στην παραγωγή ενέργειας, στην παραγωγή, μάλλον στη βιομηχανική παραγωγή χάλιβα, για παράδειγμα. Βλέπετε εδώ τώρα ένα, ένα γράφημα, ένα, ένα πίνακα που είναι πολύ ε, περίπλοκος. Το μπλε είναι το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Το κίτρινο είναι το δίκτυο μεταφοράς αερίου. Για να μπορέσουν να συνδυαστούν και τα δύο, Χρειάζεται κάτι άλλο που είναι η τεχνολογία του υδρογόνου. που θα βοηθήσει το περιορισμένο σύστημα, το περιορισμένο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας δηλαδή, να γίνει ισχυρότερο τα χρησιμοποιώντας το δίκτυο της μεταφοράς και διανομής αερίου. Ε, για το μέλλον έχετε 8 σενάρια, καθένα από αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο. Το, εκεί το υδρογόνο παίζει σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά. Υπάρχει και το ηλεκτρικό σενάριο, αλλά πρέπει να αναπτυχθεί πολύ το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και αυτό δεν συμβαίνει. Άρα είναι πιθανότερο να αποανθρακοποιηθεί το δίκτυο διανομής αερίου. Η μελέτη McKenzie που δημοσιεύθηκε πρόσφατα για την Ευρώπη δείχνει ότι εάν ακολουθήσουμε τον δρόμο του υδρογόνου μπορούμε να φτάσουμε σε μείωση κατά 560 του διοξιδίου του άνθρακος ανά χρόνο, 24, δηλαδή σχεδόν το 1 τέταρτο της τελικής ενέργειας, ζήτησης ενέργειας βασισμένη στο υδρογόνο, τα ε, έσοδα από το υδρογόνο θα είναι της τάξης των 820 δισεκατομμυρίων τον χρόνο, μείωση των τοπικών εκπομπών οξυδίου του αζότου κατά 15% και αύξηση των θέσεων απασχόληση κατά 5,4 εκατομμύρια στου σχετικού τομεί. Και όλα αυτά μέχρι το 2050. Η μελέτη αυτή είναι νοπή. Θα δημοσιευτεί σύντομα στη ε, διάσκεψη των Υπουργών Ενέργειας στο Βουκουρέστι. Αν θέλετε όμως μπορείτε να τα βρείτε στην FCHU στην ιστοσελίδα δηλαδή τη Ένωση για το Εδρογόνο. Εδώ βλέπετε διάφορε εφαρμογέ που αναμένουμε να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Βλέπετε μικρά τρίγωνα που δείχνουν την διείσδυση στις ε, μαζικές αγορές. Θα δείτε ότι για τις περισσότερες εφαρμογές για την κινητικότητα αναμένονται αυτές οι διεισδύσεις τα επόμενα 7 χρόνια. Χάρη στις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευχαριστώ πάρα πολύ και όσους συμμετέσχετε χθε στον τριμερή διάλογο, διότι είναι πάρα πολύ σημαντική η προσπάθεια αυτή, ασκούν πίεση και βεβαίως τα αυτοκίνητα που κινούνται με υδρογόνο είναι πάρα πολύ σημαντικά για την υπόθεση αυτή. Δεν θα μπω σε όλες τι τεχνολογίες τώρα. Αν δείτε περισσότερες καινοτόμες πηγές ενέργειας και ε, μάλλον ε, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, θα δείτε ότι θα υπάρχει και περισσότερο υδρογόνο, διότι είναι αναγκαίε οι πηγέ αυτέ ενέργεια. Και έρχομαι τώρα στο θέμα τη αποθήκευση. εφόσον θα έχουμε περισσότερε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, χρειαζόμαστε και μεγαλύτερου χώρου αποθήκευση. Τα είπαμε αυτά. Είναι σημαντικό να κατανοήσει κανεί ότι θα έχουμε δυνατότητε αποθήκευση εφόσον χρησιμοποιούμε υδρογόνο. 36 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μπορούν να χωρέσουν στο δίκτυο διανομής αερίου. Το ίδιο θα ισχύσει για το υδρογόνο, με 40 ε, τεραβατόρες υδρογόνου. ...18 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ε, ορυχείων άλατος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δέσμευση και αποθήκευση υδρογόνου. Είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένο το δίκτυο διανομή αερίου παντού. Τώρα, από πού να αρχίσει κανείς, από πού βρίσκεται σήμερα το υδρογόνο. Είναι τη τάξη του 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ ως, ε, ε, ο κύκλος εργασιών ανά έτος. Χρησιμοποιείται στην Ευρώπη κυρίως ε, στην μεταποίηση, βέβαια η αμμονία που χρησιμοποιείται για τα λιπάσματα, η μεθανόλη και άλλα χημικά λιγότερο σημαντικά εν τέλει και χρησιμοποιούνται συνολικώς 325 ε, μεγαβατόρες ε, υδρογόνου. Θα δείτε τώρα τι γίνεται στον πίνακα αυτό με την χημική παραγωγή αμμονίας, μεθανόλης κλπ. καθώς και την ε, σύλληψη και αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακος, CCU, θα δείτε ε, στην γαλάζια στήλη που έχετε κάτω-κάτω τον χάλιβα. Μέχρι το 2050, 390 πέτα τζάουλ, το οποίο είναι τεράστιο, τεράστια ποσότητα ενέργειας. Ε, προηγουμένως μίλησε ένας Ολλανδός ομιλητής. Εδώ βλέπετε τώρα ένα πίνακα, χάσνη, Τη εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής αερίου στην Ολλανδία αλλά και σε ένα μέρος της Γερμανίας και αυτός είναι ο δικός χάρτη που επιθυμεί να υλοποιήσει η, σχετική, η συγκεκριμένη αυτή η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται προετοιμάζεται τώρα η δέσμη μέτρων για το αέριο, ε, για, θα τα κάνει αυτά η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει νόημα να κοιτάξει τάση κανεί τη διαφάνεια αυτή, διότι οι Ολλανδοί είναι πολύ υπερήφανοι για την εταιρεία του αυτή και τα εφαρμόζουν τα πράγματα αυτά. Δεν πρόκειται απλώ για όραμα, είναι σχέδιο το οποίο θα υλοποιηθεί. Μεταξύ αυτών και αιωλική ενέργεια offshore που χρησιμοποιείται για την ηλεκτρόληση και για την παραγωγή υδρογόνου και βέβαια θα πρέπει το αέριο να αντικατασταθεί από κάτι άλλο στην ε, Ολλανδία, διότι το φυσικό αέριο έχει προκαλέσει και σεισμικές δονήσεις στο βορρά της ε, Ολλανδίας και θα πρέπει να αντικατασταθεί από το υδρογόνο. Βλέπετε εδώ μια διαφάνεια που δείχνει ότι η χρήση του υδρογόνου γίνεται πλέον εμπορικά σημαντική. Άλλο Ολλανδικό παράδειγμα του λιμανιού του Άμστερνταμ με Νουριόν, Τάτα Στυλ και Αξονομπέλ που ε, χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες αυτές αλλού σε δηληστήριο που χρησιμοποιεί την ηλεκτρολύση όχι μόνο για να δημιουργήσει, να παραγάγει μάλλον υδρογόνο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί μετά για την ε, παραγωγή χάλιβα, αλλά και το διαθέτουν και στα δίκτυα διανομής. Και έχετε επίσης και το H2 Future, αυστριακό, μιλήσαμε και για τη Σουηδία, μιλήσαμε για τη Γερμανία, δεν μιλήσαμε για το ThyssenKrupp, όπου ο νέος τους διευθυντής μίλησε, είπε ότι τον Απρίλιο θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν ε, τεχνολογίες σύλληψης και αποθήκευσης του διοξιδίου του άνθρακος για να φτάσουν μέχρι το 2050. Αυτά ήταν η δική μου παρουσίαση και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για, για την παρουσίασή σας. Ξεκινάει τώρα η συζήτηση. Έχετε το λόγο, κύριε Γκύρα. E, σας ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι πώς ακριβώς μπορούμε να αποθηκεύσουμε το υδρογόνο. Το υδρογόνο παρουσιάζει κάποια χαρακτηριστικά ιδιαίτερα επικίνδυνα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο μπορούμε να προστατευθούμε από πιθανά ατυχήματα του υδρογόνου. Ξέρετε ότι είναι διασπόμενο εύκολα και συνεπώς επικίνδυνο. Πώς μπορούμε να προστατευθούμε. Έχουμε δύο τεχνολογίες για την παραγωγή υδρογόνου. Η μία είναι η ηλεκτρόλυση και η άλλη είναι η παραγωγή από τον άνθρακα. Η αποτελεσματική ε, χρήση της ενέργειας ε, πού επιτυγχάνεται, ποια είναι η καλύτερη τεχνολογία για το μέλλον. Παρακαλώ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Να υπογραμμίσω ότι φυσικά Προσπαθούμε να προσαρμόσουμε την προσοχή μας στα θέματα του υδρογόνου. Αλλά όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε γενικότερα την χρήση των αερίων στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι στην ουσία έχουμε να κάνουμε με μια ανάμιξη προϊόντων από διαφορετικές πηγές. Θα μπορούσατε λοιπόν να αναλύσετε λίγο ακριβώς πώς ε, θα μπορούσε το υδρογόνο να αναμειχθεί με άλλα αέρια και να μεταφέρεται με σωληνώσεις για οικιακή χρήση ας πούμε. Και ποια είναι η επιπλέον πηγή και η επιπλέον τεχνολογία η οποία θα μπορούσε να το παράγει. Ε, εδώ τίθεται το θέμα και της βιομηχανίας βιοαερίων και τι ορισμοί χρησιμοποιούνται, πράσινο αέριο, μη χρήση άνθρακα. Ε, θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι λοιπόν και να μην έχουμε όρους οι οποίοι είναι γενικότερα γενικόλογοι και θολοί. Δεύτερον, ο κύριος Γκέρεκ είπε ότι για το υδρογόνο υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής και από άνθρακα. Λαμβάνοντας υπόψη και την προηγούμενη παρατήρησή μου, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο παράγεται το υδρογόνο. Δεν θα πετούνται συγκεκριμένα ισχυρά κριτήρια βιωσιμότητας γιατί το υδρογόνο θα μπορούσε να είναι ένας καλός τομέας για την ενεργειακή μετάβαση, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί αυτό σκοπό. Έχει ένα ρόλο να παίξει λοιπόν στην ανθρακοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας, το στηρίζω αυτό, αλλά δεν είναι, επαναλαμβάνω, ένας αυτός σκοπός η χρήση περισσότερου υδρογόνου στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Νομίζω λοιπόν ότι μια ε, απαιτούνται αυστηρότερα κριτήρια βιωσιμότητας για το υδρογόνο από ό,τι για τα υπόλοιπα αέρια. Και μια τρίτη ερώτηση είναι κάτι σχολιάσατε ιδιαίτερα για την αποθήκευση του υδρογόνου. Το θέμα είναι και οι κανονισμοί που θα διέπουν τα δίκτυα, τη λειτουργία των δικτύων. Πώς εσείς φαντάζεστε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος, το υδρογόνο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αποκλειστικά με βάση την αποθήκευσή του, αλλά και της, ε, την ευκολία μετακίνησης, ε, την ένταξή του στα δίκτυα. Αυτό θα μειώσει το κόστος πιθανώς. Ο κύριος Έλα. Να επανέλθω στην εργασία μας. Είχαμε αυτό το Hydrogen Undertaking, το οποίο υποστηρίξαμε στον ορίζοντα 2020. Τώρα, mm το ιστορικό επιτυχίας του Hydrogen Undertaking είναι δύσκολος. Δύσκολο, διότι η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα και προβλήματα κόστους και της έφυγε λίγο η διάθεση να ασχοληθεί με το υδρογόνο. Βλέπει τώρα προφανώς ότι αντιμετωπίζει προβλήματα με τους συσσωρευτές και το ξανασκέπτεται. Τώρα, σχετικά με μια μελλοντική κοινοπραξία υδρογόνου, τι στόχους θα πρέπει να έχει και σε, ποιο, σε ποιες τάξεις μεγέθους ώστε να συνεργαστεί η βιομηχανία. για να φτιαχτεί ένα hydrogen, hydrogen joint undertaking νούμερο 2 ή και νούμερο 3 ενδεχομένως το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντικό να σκέπτεται κανείς το μέλλον. Απαντήσεις. Να αρχίσω με τις πρώτες και να αφήσω τις δύσκολες για το Χατζημαρκάκι. Πρώτα λοιπόν, πρώτη ερώτηση ήταν σχετικά με το ότι είναι ασταθές και επικίνδυνο αέριο το υδρογόνο. Έχουμε μεγάλη εμπειρία με 3.000 χιλιόμετρα αγωγών υδρογόνου που η πρώτη φτιάχτηκε το 1938 και συνεχίσει να λειτουργεί, το υδρογόνο είναι επικίνδυνο με διαφορετικό τρόπο από το φυσικό αέριο. Δεν είναι συγκρίσιμα δηλαδή από την άποψη της ασφάλειας. Υπάρχουν άλλοι που μιλούν για την ασφάλεια και λένε ότι το υδρογόνο δεν είναι λιγότερο επικίνδυνο από το φυσικό αέριο, αλλά είναι διαφορετική κίνδυνη. Βέβαια υπάρχει και το διοξείδιο του άνθρακο ή το οξύδιο του άνθρακο το οποίο μεταφέρεται με αγωγού. Για την παραγωγή τώρα του υδρογόνου μπορεί να προκύψει και από την βιομάζα. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί θα μείωνε και τι ε, εκπομπέ. Μια ερώτηση τέθηκε σχετικά με την ανάμιξη υδρογόνου στο φυσικό αέριο πολλοί έχουν πιέσει για να ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δίκτυα μεταφοράς του φυσικού αερίου. Πριν από μερικά χρόνια, ωστόσο, οι εταιρείε που ε, διοχετεύουν φυσικό αέριο δεν σκέπτονταν τα σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων μέχρι που τις υποχρέωσαν οι κυβερνήσεις. Τώρα, δεν θα είναι καλή επιλογή αφού δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει σε διοχέτευση πάνω από 20% υδρογόνου και ίσως χαμηλότερο πάντως, όχι πέρα από 20%, γιατί δίθεται και θέματα ταχύτητας μεταφοράς του υδρογόνου κλπ. Αν θέλετε να χρησιμοποιηθεί το υδρογόνο στα δίκτυα διανομής του φυσικού αερίου, θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλές αλλαγές. Μπορώ να πω πάντως ότι αν θέλετε να περάσετε από αυτή την μετατροπή, οι περισσότερες μετατροπές θα πρέπει να γίνουν στα, στις συσκευές τελικής χρήσης του αερίου και όχι στο ίδιο το δίκτυο. Για την ε, βιωσιμότητα του υδρογόνου. Δεν πρόλαβα να σας δείξω την τελευταία μου διαφάνεια γιατί έληξε ο χρόνος μου. Η ορολογία που χρησιμοποιούν είναι πράσινο υδρογόνο, χαμηλά, χαμηλός άνθρακας κλπ. Προτείνονται διάφορα πρότυπα για τη χρήση του υδρογόνου και τα πιο προηγμένα και πιο πρόσφατα είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο πρόβλημα είχαν, είχε και το ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να αρχίσουμε πρώτα με την ανάμιξη. Ναι, έχει νόημα η ανάμιξη μέχρι 20% για τη μεταβατική περίοδο. Μετά από 20% μπαίνει θέμα. Χρειάζεται να αλλάξουν και η αγωγή αλλά και οι συσκευές των καταναλωτών. Ίσως έχει όμως νόημα για το μέλλον ε, χρειάζονται ειδική αγωγή, αλλά είναι τόσο ε, τέτοιε διαμέτρου. Ε, αυτές που υπάρχουν μάλλον είναι τόσο μικρές που σας δείχνω, δηλαδή τη των 12 εκατοστών διαμέτρου, αλλά θα χρειαστούν ε, πολύ ε, μεγαλύτερη, ας πούμε του μισού μέτρου. Ακούσατε ποτέ για κανένα ατύχημα, όχι, γιατί έχουμε υψηλά επίπεδα ασφαλείας, υψηλά πρότυπα ασφαλείας. Ακόμα και για τις ε, στοές όπου φυλάσσεται το υδρογόνο, ακόμα και τι είδους βακτήρια επιτρέπεται να υπάρχουν μέσα εκεί. Θα ήθελα τώρα να απαντήσω στην ερώτησή σας για τους διάφορους τρόπους παραγωγής του υδρογόνου. Πράγματι, από ατμούς μεθανίου, από φυσικό αέριο ή από άνθρακα, η αεριοποίηση του άνθρακα δηλαδή, 95% του σημερινού υδρογόνου προέρχεται από εκεί. Αν προχωρήσετε στο CCS, τότε γίνεται η αποανθρακοποίηση. Υπάρχει και η ηλεκτρόλυση η οποία ενισχύεται. Το 80% βέβαια, αν πάτε στην ηλεκτρόλυση, είναι το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματο που χρησιμοποιείται για την ηλεκτρόλυση. Υπάρχει και μια τρίτη επιλογή, η τεχνολογία η οποία ξεκίνησε από τη γερμανική BASF και την εξετάζει και η ε, Gazprom και είναι η πυρόληση. Η πυρόληση είναι τρόπος παραγωγής, παραγωγής υδρογόνου και σταθερού άνθρακα υπομορφή ε, σκόνης. Αυτή η σκόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να, ε, ως πρώτη ύλη, για παράδειγμα για ελαστικά αυτοκινήτων, ως γραφίτης ή μπορεί να το θάψει κανείς. Εγώ προέρχομαι από το Σάρλαντ, όπου σταματήσαμε την εξόριξη του άνθρακα και αυτό που θα μπορούσε να κάνει κανείς θα ήταν να γεμίσει τις στοές των ορυχείων με, με αυτή την σκόνη και να τη θάψει εκεί μέσα. Τότε θα έχετε υδρογόνο. Ε, εξετάζουμε τώρα πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό και αν το επιτρέπουν και οι τιμές. Τα είπε η BASF αυτά πριν από λίγο καιρό. Διότι η πυρόληση είναι 10 φορές φθηνότερη από την ηλεκτρόληση. Αυτό ήταν νέο στοιχείο για μένα, το ομολογώ και το εξετάζουμε, το σωστό ομολογώ, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την Πολωνία συγκεκριμένα τώρα. JSW, η μεγαλύτερη ε, επιχείρηση εξόριξης άνθρακα που ε, ζήτησε να γίνει μέλος μας, όχι για να φτιάξουμε από τον άνθρακά τους υδρογόνο, αλλά διότι θέλουν να σταματήσουν την παραγωγή του άνθρακα και θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα ορυχεία που έχουν εξαντληθεί για χρησιμοποίηση ε, ε, να χρησιμοποιηθούν για, τη, για τα ε, υπόλοιπα της ηλεκτρόλυσης. Και επανέρχομαι στον κύριο Έλερ. 40 δισεκατομμύρια τώρα θα διαθέσει η Γερμανία για τη μεταβατική περίοδο. Χρήματα. Εμεί βρισκόμαστε ήδη σε συνομιλίε με τα Υπουργεία και τα Περιφερειακά Υπουργεία Ενέργειας τη Γερμανία για τις επενδύσεις για την τεχνολογία παραγωγής. Και να μην, να μην πάνε τα λεφτά αυτά τελικά στην Κίνα. Είπαν οι κυβερνήσει ότι θα φτιάξουν και μια μονάδα. Γιατί εμείς ε, έχουμε λάβει τον τίτλο IPCI, δηλαδή ε, έργο που είναι σημαντικό για την ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγή. Χρειαζόμαστε 4 γιγαβάτ τον χρόνο για την ηλεκτρόληση. Θα δούμε, θα πάμε στο Αμβούργο, θα πάμε στη Βόρεια Ιρλανδία, Βεσσαλία, στην Ισπανία, στην Πολωνία και θα προχωρήσουμε με τα σχέδια αυτά βιομηχανοποίηση. Να απαντήσω στην ερώτησή σου τώρα για την κοινοπραξία. Πράγματι, η κοινοπραξία βασίστηκε ιδίω στην μεταφορά. Στι μεταφορέ, μάλλον. Χρήση δηλαδή καθαρού υδρογόνου σε αυτοκίνητα. Και πράγματι, κάπου έχουμε σημεία εχμή. Πολλέ χώρε μέλη, η Γερμανία για παράδειγμα, έχει 56 σταθμού ανεφοδιασμού, δεν έχει όμω αρκετά αυτοκίνητα που να κινούνται με υδρογόνο. Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Διότι τα γερμανικά ΟΕΜ, και μιλώ για τα μέλη μου, είναι, ε, καθυστερούν πολύ. Όμω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει ένα ρόλο. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει διαρκώ μόνο το ένα μοναδικό μήνυμα ε, επικεντρωθείτε στου συσσωρευτέ, δηλαδή ηλεκτρικού συσσωρευτέ, ε, τότε δεν θα πάει, δεν θα προχωρήσει το υδρογόνο. Είμαστε βέβαιοι λοιπόν ότι το υδρογόνο στα αυτοκίνητα θα τεθεί ω θέμα, διότι είναι βολικό και είναι μια τεχνολογία όρημη Όμως το κοινό συζητεί ιδίω για συσσωρευτέ. Και χρειάστηκε χρόνος βέβαια για να φτάσουμε εκεί. Τώρα το μελλοντικό, η μελλοντική κοινοπραξία δεν θα πρέπει να περιοριστεί στις μεταφορές. Και γι' αυτό είναι τόσο συναρπαστικό ε, για μένα που εργάζομαι σε αυτόν τον κλάδο. Είναι για, πρόκειται δηλαδή για την συγκέντρωση των τομέων, των κλάδων, sectoral integration, ώστε τα συστήματα αυτά να συνεργαστούν μεταξύ τους για να φτιάξουν τα σωστά σημεία διατομής μεταξύ ηλεκτρικών δικτύων και δικτύων αερίου. Και χρειάζεται να γίνει αυτό και θα το χρειαστούμε περισσότερο στο μέλλον. Εάν στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση ρίξει το βάρος της μονάχα σε ένα, ας πούμε μόνο στο χάλιβα ή μόνο στις μεταφορές, θα αποτύχει να κατανοήσει ότι το υδρογόνο είναι τεχνολογία κλειδί για να λειτουργήσουν αυτά τα σημεία διατομής, interfaces, για να μεταφέρει την ε, ε, ανανεώσιμη ενέργεια στις μεταφορές, στην θέρμανση των κατοικιών και ούτε καθεξής. Είμαι ανοιχτό μαζί σου, Κρίστιαν, γιατί εσύ έπαιξε σημαντικό ρόλο και είναι δύσκολο να βρει κανεί κάποιον που να γνωρίζει το ορίζον Ευρώπη τόσο καλά και μπόρεσε και έριξε μια καθαρή ματιά σε αυτό. Το ξέρω. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Τα σημεία εχμή βρίσκονται σε ορισμένε χώρε μέλη, όπω πάντα. Μπορώ να σα πω όμω ότι για δεύτερη φορά Τώρα, οι Υπουργοί ενέργεια έχουν βάλει το υδρογόνο ως θέμα τους. Στο Λίντεν τη Αυστρίας, την τελευταία φορά δηλαδή που συνειδήθηκαν άτυπα και το συζήτησαν, την επόμενη φορά θα συναντηθούν στο Βουκουρέστι. Δεν παραπονούμεθα. Οι Υπουργοί είναι ανοιχτοί για να το συζητήσουν το θέμα αυτό, αλλά πρέπει να κινηθούν ταχύτερα, διότι η Κίνα και η Ασία γενικότερα είναι πολύ ταχύτερες από εμάς για την ώρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους δύο καθηγητές για τις ε, απαντήσεις σας, για όλες τις πληροφορίες. Ήταν πολύ χρήσιμο. Είχαμε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ πρόσφατα και εκπροσώπους από την, το Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων. Πολύ σημαντικός οργανισμός. Και δεν χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά την κουβέντα υδρογόνο. Εγώ τους έθεσα την ερώτηση γιατί είναι σημαντικό το θέμα. Και η απάντησή τους ήταν με λίγα λόγια είναι ανανεώσιμες ως πρωτογενής ενέργεια, ως, ως πηγή πρωτογενούς ενέργειας. Το υδρογόνο είναι άλλο. Διότι δεν έχουμε καθαρό υδρογόνο στη φύση. Από αυτή λοιπόν την πλευρά είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για όλες τις εξηγήσεις σας και τις εισηγήσεις. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, πιο απλά τα μάλλον τα πράγματα, ανανεώσιμες και πράσινες λύσεις, ίσως και λίγο αέριο. Αλλά αυτό πρέπει να εισάγουμε από την ε, σκοπιά και τη διάσταση των στρογών πρέπει να πάει προς τις ανανεώσιμες. Αυτό θα ήταν χρήσιμο για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ και τελευταίο μέρος του πάνελ μας. Τρίτο πάνελ, παράδειγμα της ενεργειακής μετάβασης στη Γερμανία. Ο Ραφάου Μπάτσουκ. Ε, συνεργάτης, ε, καθηγητής στο κέντρο για τις ανατολικές μελέτες, ειδικό ε, για τα θέματα των κλιματικών αλλαγών στη Γερμανία. Και το θέμα μας είναι ακριβώς αυτό, η μετάβαση προς την παραγωγή ηλεκτρισμού χωρίς άνθρακα στη Γερμανία. Και μετά η οικονομία της Γερμανίας γενικότερα ως προς την ενέργεια, με τελευταία δημοσίευση η γερμανική ενεργειακή πολιτική και το αβέβαιο του άνθρακος και της βιομηχανίας που βασίζεται σε αυτόν στη Γερμανία. Συναρπαστικότατο. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Σε ποια γλώσσα, αγγλικά, γίνεται. Good morning. good morning. Uh, I'm to speak Καλημέρα σας, είναι Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω, να εξηγήσω το Κέντρο Ανατολικών Σπουδών. Είναι ένα κυβερνητικό κέντρο ερευνών ασχολούμεθα με θέματα τα οποία άπτονται της γειτονίας στην χώρα μου, στην Πολωνία, κυρίως ε, με θέματα και στη Γερμανία. Και εγώ ασχολούμαι με τη βιομηχανική πολιτική της Γερμανίας και την ενεργειακή πολιτική, την στρατηγική εξόδου από τον άνθρακα της Γερμανίας, Πρώτα θα μιλήσω για, τα γενικότερα, ε, για τη γενικότερη κατάσταση στον τομέα της ενέργειας. Είναι μια μακροπρόθεσμη προοπτική η ενεργειακή πολιτική της Γερμανίας. Στόχος είναι η απομάκρυνση από τον άνθρακα. Το 2050 θα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές κατά 80 με 95%. Να αυξηθεί υποτίθεται η χρήση των εναλλακτικών πηγών Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Όταν βλέπουμε εδώ τις κίτρινες ετικέτες, βλέπουμε ότι η στρατηγική αφορά την καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη. Δεν είναι μόνο απλά ενεργειακή πολιτική, αλλά γενικότερα οικονομική στρατηγική της χώρας και υπάρχει μια συναντήληψη στους Γερμανούς πολιτικούς και τη γερμανική βιομηχανία ότι υπάρχει ανάγκη για μεταρρύθμιση της γερμανικής βιομηχανίας και των τρόπων με τον οποίο επιτυγχάνει τους στόχους. Τώρα πώς επιτυγχάνει ακριβώς τους συγκεκριμένους στόχους βλέπουμε στο γράφημα εδώ ότι βασικός στόχος είναι το 2050 η επίτευξη του 80% μείωσης. Η πράσινη γραμμή εδώ διαφέρει όπως βλέπετε ήδη από το 2018. Φτάσαμε περίπου στο 40%. Έχει ξεπεραστεί ο αρχικός στόχος όταν βλέπουμε ε, γενικότερα το θέμα της εκπομπής ε, αερίων. Εδώ η Γερμανία δεν έχει ακόμα καταφέρει να πετύχει τους στόχους. Η κυβέρνηση είπε, ε, είπε ότι δεν θα πετύχει το 40% το 2020, όμως Υποτίθεται ότι προσπαθεί να πετύχει πάντα τον στόχο του 55% για το 2030. Το 2018 η κυβέρνηση ε, πέρασε ένα νόμο για θέματα κλιματολογικών ε, αλλαγών και αυτό αφορά και στην παραγωγή εκπομπών από την ε, ηλεκτρική ενέργεια εδώ βλέπετε την ηλεκτρική ενέργεια, την ενέργεια από τα ορυκτά καύσιμα και την ενέργεια από τον άνθρακα. Ο άνθρακας παράγει το 40% του, της ενέργειας. Τώρα για την έξοδο από τον άνθρακα δεν υπάρχει μια πλήρη στρατηγική ακόμα, υπάρχει όμως μια πολιτική ε, συνένεση θα έλεγα για να υπάρξει αυτή η πραγματική έξοδος. Έχουν γίνει συζητήσεις ανάμεσα στους εκπροσώπους της κυβέρνησης και τα λόμπι των βιομηχανιών. Έγιναν ήδη ορισμένε κοινέ προτάσεις. Βλέπουμε τις προτάσεις αυτές στη χάρτα. Βλέπετε ότι το 2025 με 2030 ε, ε, οι μονάδες παραγωγής ε, με άνθρακα οι περισσότερες θα σταματήσουν την παραγωγή τους, θα απαιτηθούν επεμβάσεις από τα διαφθρωτικά ταμεία σε περιφέρειες οι οποίες εξαρτώνται σε ένα μεγάλο βαθμό από την εξαγωγή και την χρήση του άνθρακα, πώς θα γίνει αντικείμενο διαχείρισης η μεταπατική περίοδος που θα ακολουθήσει το κόστος του προγράμματος θα είναι περίπου 40 δις τα επόμενα 20 χρόνια. Όπως είπα στο παρελθόν, η έξοδος από τον άνθρακα δεν είναι κάτι το οποίο έχει καθοριστεί ε, με νομική, ε, με δεσμευτικό νομικό τρόπο. Σχετικά τώρα με το μείγμα του ηλεκτρικού, ηλεκτρικού ρεύματος βλέπουμε ότι οι ανανεώσιμες το 2035 θα φτάσουν περίπου στο 50%. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι ε, το φυσικό αέριο και αυτό θα πενταπλασιαστεί με τους αριθμούς που ίσχυαν μέχρι τώρα και θα φτάσει περίπου το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας θα παράγεται δηλαδή από το φυσικό αέριο, κάτι το οποίο θα έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις <clears throat> για τον ρόλο και το ποσοστό του φυσικού αερίου στα πλαίσια του μείγματος των ενεργειών που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η έξοδος λοιπόν από τον άνθρακα οφείλεται κυρίως στη μείωση ε, των ε, εκπομπών. Βλέπουμε στον χάρτη εδώ μπροστά ότι δεν είναι μόνο η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος που παράγει εκπομπές, δεν ξεπερνάει το 55%. Το 2030 θα υπάρξουν παρεμβάσεις και στον τομέα της οικοδομής και στον τομέα της βιομηχανικής δραστηριότητας εκτός ενέργειας και στον τομέα των μεταφορών οι μεταφορές προσφέρονται ιδιαιτέρως. Ε, γνωρίζουμε ότι στις μεταφορές υπάρχει ένα πάρα πολύ ισχυρό γερμανικό λόμπι και μέχρι τώρα δεν έχουν ακριβώς ε, ε, δηλώσει το ποια πορεία θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα. Τώρα, σε σχέση με το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, εδώ βλέπετε το κόστος από παραγωγές, από ενέργειες ε, ηλιακές, ε, ηλιακή ενέργεια, αιωλική ενέργεια. Η αύξηση του ε, ποσοστού των εναλλακτικών θα επηρεάσει θετικά το ύψος των τιμών Κάτι το οποίο όμως εδώ στα πλαίσια του γραφήματος αυτού είναι πολύ δύσκολο να ορίσει κανείς. Και θα πρέπει να δούμε εμείς και τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο πολιτικό. Ο χάρτης αυτός δείχνει τις χώρες οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει ε, την πορεία εξόδου από τον άνθρακα και χώρες οι οποίες δεν το έχουν ακόμα αποφασίσει. Βλέπετε ότι υπάρχει μια σχετικά ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή. Μια μειοψηφία των ανατολικών χωρών παραμένουν πιστές εισαγωγικά στον άνθρακα είναι σαφές ότι εδώ υπάρχει μια έλλειψη πολιτικής ενότητας ε, και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα και για τις υπόλοιπες χώρες να εμπλακούν στην οδό της απαλλαγής από τον άνθρακα. Και ο τελευταίος χάρτης εδώ δείχνει το μέγεθος στην Ευρώπη της εξαγωγής άνθρακα Πολωνία, Τσεχία, είναι χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν πάρα πολύ τον άνθρακα. Θα πρέπει να δείτε τις Βαλκανικές χώρες, τη Νότια Ευρώπη. Οι χώρες αυτές χρησιμοποιούν λιγνίτη. Δεν θα θέλαμε στο μέλλον να πηγαίνουν ε, εξοπλισμοί για την ε, παραγωγή λιγνίτη, ε, γιατί ξέρουμε ότι ο λιγνίτης δημιουργεί πάρα πολλά κλιματολογικά προβλήματα, η χρήση του λιγνίτη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα παραδείγματα που εξηγήσατε. Ευχαριστώ και για τις διαφάνειες. Τώρα ακολουθεί ο καθηγητής κύριος Χάκερ από το Ινστιτούτο Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών για αξιολόγηση τεχνολογιών και ειδικό για την ενεργειακή μετάβαση στην γερμανική οικονομία. και για την εφαρμογή συμφωνιών κλπ. Τεχνολογιών άνθρακος και τεχνολογίες μείωσης των οξυδίων του άνθρακος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ο τελευταίος λοιπόν για το σημερινό πρωινό και δεν είναι και τόσο εύκολος ο ρόλος μου διότι τα βασικά τα είπαν ήδη. Αυτό που καλούμε να κάνω είναι τώρα να συνοψίσω κάπως τη συζήτηση. Αλλά πώς. Σε κάποιο βαθμό διαμορφώνεται μια συνένεση σε ό,τι αφορά τις απόψεις μας σχετικά με το πώς θα πρέπει να μετατρέψουμε τα εθνικά μας συστήματα ενέργειας. Δηλαδή γνωρίζουμε τι απαιτείται. Έχουμε και συστήματα στόχων κατατεθειμένα στο τραπέζι που διαφέρουν από χώρα σε χώρα βεβαίως αλλά θα ήταν και βαρετός ο κόσμος αν δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ μας. Ίσως είναι και το αλάτι ας πούμε της ευρωπαϊκής μαγειρικής αυτό. Εγώ δεν θα επαναλάβω και ως καθηγητής ομολογώ ότι δεν ε, διεπίστωσα να έχει σφάλματα η παρουσίαση του νεαρού συναδέλφου μου δίπλα μου. Θα ήθελα ε, να έλθω όμως κυρίως στην τρέχουσα κατάσταση στη Γερμανία τώρα. Τα γνωρίζετε αυτά, διότι είναι αυτά που έλεγε και το θεμελιώδες εγχειρίδιο προδεκαετίες προδεκαετίας όταν είχαμε αρχίσει να μιλούμε για την ενεργειακή μετάβαση στην ε, ε, Γερμανία που τότε είχε θερμανθεί βεβαίω η συζήτηση διότι η μετατροπή αυτή ε, δεν έγινε καλά δεκτή από όλα τα στρώματα της κοινωνίας μας και παρακολουθεί το και με κάποια επιφύλαξη και καχυποψία και από τις γειτονικές χώρες. Δηλαδή σκεφτόντουσαν αυτοί οι τρελοί Γερμανοί τι έχουν αρχίσει να κάνουν πάλι τώρα. Εάν θέλει κανείς να τα αναλύσει, η βασική προτεραιότητα είναι η μείωση από όλους τους τομείς των εκπεμπόμενων οξυδίων του άνθρακος. Αυτός ο στόχος εξαφανίζεται. Αν, αν μάλλον ο στόχος αυτός εξαφανιστεί, θα έχει σημαντικότατη επιρροή στις μελλοντικούς, στους σχεδιασμούς. Αυτό δηλαδή που θα πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι, είναι ότι όλες οι σχετικές στρατηγικές, οράματα κλπ ξεκινούν από αυτή τη σημαντική προτεραιότητα κλειδί στη χώρα μου. Έχετε δει ήδη τα δεδομένα. Βρισκόμαστε τώρα στην συζήτηση μετά από την πολύ καυτή συζήτηση για τον περιορισμό της πυρηνικής ενέργειας, μιλούμε τώρα για τη σταδιακή μείωση και κατάργηση του άνθρακα. Και θα είναι πολύ δύσκολη επιλογή. Ακούσατε ορισμένα πράγματα που είναι δυνατόν να γίνουν, αλλού που δεν είναι και ως ε, κάπως πιο ε, ηλικιωμένος πανεπιστημιακός οφείλω να σας πω ότι έχω ακούσει τόσα παραμύθια για το μέλλον της Γερμανίας και τα μελλοντικά συστήματα ενέργειας όταν ακούω ότι φτάνουμε σύντομα στην καταστροφή και ποτέ δεν θα μπορέσουμε να τα πετύχουμε όλα αυτά τα πράγματα τότε κλείνω τα αυτιά μου συνήθως διότι τις περισσότερες περιπτώσεις δεν αξίζει καν τον κόπο να ασχοληθεί κανείς με τα σενάρια αυτά. Το μείζον θέμα, όταν συζητούμε αυτή τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα, στρέφεται κυρίως γύρω από το μέλλον του λιγνίτη στην Γερμανία. Και το ερώτημα είναι τι είδους διαρθρωτική αλλαγή θα προκληθεί στις περιφέρειες ιδίως που τον παράγουν. Και μιλώ για απασχόληση. Και την τονίζω τρει φορέ. Απασχόληση, απασχόληση, απασχόληση. Και τελικώ πρόκειται για χρήματα. Με λίγα λόγια δηλαδή, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως τώρα για αυτή την ενεργική μετάβαση στην Γερμανία είναι ότι αφενός μειώνουμε το χαρτοφυλάκιο, το τεχνολογικό μας χαρτοφυλάκιο και αυξάνουμε την, ε, τις επιλογές. Από την άλλη μεριά αυτό κάτι που συζητείται πολύ είναι ότι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια όλο και μεγαλύτερη αστάθεια, ιδίως για την παροχή ενέργειας σε αστικά κέντρα. Για την αποθήκευση, για παράδειγμα, του, των οξυδιών του ανθρακός. Είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε καταφέρει ως τώρα να χειριστούμε καλά αυτή την αστάθεια. Βεβαίως μας περιμένουν προκλήσεις. Προσωπικά από τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου δεν φοβούμε τόσο πολύ την αστάθεια αυτή διότι μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε εάν προχωρήσουμε με ε, λογικό τρόπο. Εάν αφήσουμε να καθοριστούν οι μελλοντικέ μας στρατηγικές περισσότερο από τα συναισθήματα τότε δεν θα πετύχουμε. Αν όμως βασιστούμε σε στέρεες τεχνολογίες και οι τεχνολογίες υπάρχουν τότε όπως είπα δεν φοβούμε το μέλλον ούτε ή οδήποτε blackout. Αντιμετωπίζουμε δυσχέρειες επίσης ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση των δικτύων. Μου ζήτησαν κύριε Πρόεδρε να μιλώ αργά γιατί το ζήτησαν υποτίθεται οι διερμηνείς. Και ο διερμηνέας σημειώνει και πολύ καλά κάνει ο κύριος Χάκε και μιλά αργά θα, ναι, θα μας φύγουν κάποιες μη διερμηνείς, λέει ο πρόεδρος, και θα μείνουν μόνο με τα αγγλικά. Έχω καλύψει 6 λεπτά ως τώρα. Η αναδιάρθρωση του δικτύου λοιπόν αποτελεί μια πρόκληση ή των δικτύων. Εκεί έχουμε δει πολλές καθυστερήσεις. Είμαστε αρκετά πίσω. Βεβαίως διεξάγεται συζήτηση για το κόστος ο κόσμος ε, δεν του αρέσει να βλέπει κοντά στο σπίτι του, δηλαδή στην αυλή του, τι ανεμογεννήτριε. Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Καλύψαμε σήμερα και τον τομέα του τελικού χρήστη, όπου έχουμε πολλά project για να δούμε πώς μπορεί να αυξηθεί η αποδοτικότητα της ενέργειας, ε, μείωση των διοξιδιών του άνθρακος κτλ. Κάτι που δεν αναφέρθηκε σήμερα το πρωί, ωστόσο, είναι και το ζήτημα της αποδοχής από πλευράς του κοινού. Εάν ακόμη δηλαδή υπάρχει πράγματι ακόμα μεγάλη ευρύτατη στήριξη για την ε, ε, ενεργή βέντε αυτή την αλλαγή, δηλαδή του, του, υποδείγματος στην ενέργεια, ε, υπάρχει ακόμα και πάρα πολλή αντίσταση ε, τοπικά απέναντι σε ορισμένες πηγές ανανεώσιμων πηγές, πηγές ενέργειας. Τώρα υπάρχει και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία υπέβαλε στις κυβερνήσεις. Διεξάγεται συζήτηση τώρα σχετικά με το σε ποιον βαθμό θα πρέπει να γίνει επίσημη ενεργειακή πολιτική της χώρας μας. Με λίγα λόγια, αυτό που βλέπουμε ως πρώτες αντιδράσεις στην έκθεση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι διεξάγεται συζήτηση για τους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων μερών που δεν ήταν και μέλη της Επιτροπής. Εννοεί μάλλον την Επιτροπή Άνθρακος ο η Γερμανική Επιτροπή Άνθρακος. Η ερώτηση που θέτουν οι Γερμανοί βουλευτές είναι, εθνικοί βουλευτές δηλαδή, πώς εμπλέκεται το Γερμανικό Κοινοβούλιο ή πρόκειται για ένα είδος αγνόησής του από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση που δεν λαμβάνει υπόψη δηλαδή τι αποφάσεις του. Ο προηγούμενος ομιλητής αναφέρθηκε ήδη και στις χρηματοδοτικές δεσμεύσει. Αυτά τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι βέβαιο να έχουν μια στέρεα βάση. Κάτι άλλο που δεν είναι τόσο σαφές είναι ποιος είναι ο απότερος στόχος για τη στρατηγική αυτή αλλαγή. Θεωρώ ότι υπερβάλλουμε σε ό,τι αφορά τη στόχευση για την ενεργειακή μεταβολή. Το ζήτημα είναι πόσο θα, πόσο θα πρέπει να μετατρέψουμε την οικονομία μας, της, της, την απασχόληση και ποιες είναι προοπτικές σε άλλους τομείς που έχουν ενδιαφέρον για την κοινωνία. Διότι αν δεν το επιτύχουμε αυτό, δεν θα έχουμε την υποστήριξη του κοινού για την ενεργειακή μετάβαση στο μέλλον. Νομίζω τα διαβάζετε αυτά και εσείς. Το μόνο που θέλω να τονίσω είναι κάτι ακόμη. Όταν σταδιακά καταργήσουμε τον άνθρακα. Έχει αρχίσει τώρα η συζήτηση και για τον αγωγό νούμερο 2 των βαλτικών χωρών. Διότι πολλοί φοβούνται ότι θα υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στις ανανεώσιμες ενέργειες και στον άνθρακα που θα έχει απομείνει. Και διερωτώνται διάφοροι μπορεί να, να, καλυφθεί το κενό αυτό με το φυσικό αέριο. Και με τη χρήση βέβαια αυτού του σημαντικού αγωγού 2. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά και από την άποψη ολόκληρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Ευχαριστώ τους διερμηνείς. Μπορούμε να έχουμε μία ερώτηση από τα πολωνικά. Μία όμως. Τελευταία, ακροτελεύθερα. Και μετά στα αγγλικά όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τη δυνατότητα. Ήθελα απλώ να μου πείτε εάν η απαλλαγή από τον άνθρακα μπορεί να αφορά και τις, τα εργοστάσια ηλεκτρικής θέρμανσης. Ξέρουμε ότι κοντά στο Αμβούργο έχει χτιστεί πρόσφατα ένα νέο εργοστάσιο, ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού. Πρώτη ερώτηση και δεύτερη, αυτή η μετάβαση προς το αέριο. Εάν το Nord Stream 2 αλλάξει τις αναλογές που αναφέρατε, 40 προς 60, θα γίνει το ανάποδο. Όμως, Όλα αυτά θα ισχύουν και για τι ίδιε τι τουρμπίνε, τι τις ε, που θα κινούνται με αέριο ή και την παραγωγή με ατμό. Ευχαριστώ πολύ όλους τους διερμηνείς. Θα ξαναβρεθούμε σε δύο ώρες στις 2.30 στην Επιτροπή Ήτρε και τώρα μπορούμε να κάνουμε τις ερωτήσεις μας αλλά θα συζητήσουμε στα αγγλικά. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. I mean, I'm, I'm